Sorry? Good morning to you. Καλημέρα σας. Επιτροπή Προπολογισμού. Σημερινή συνεδρίαση. Πρώτο σημείο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν εφαντηρήσεων εγκρίνεται. Καταρχάς, να πω ότι έχουμε δει δικαιωμένου φιλοξενούμενους στην Επιτροπή προπολογισμού. Πρώτα απ' όλα, τον αντιπρόεδρο τη κυβερνήση και υπουργό οικονομικών, Ζάφκο Μάλιτς, από την Κροατία και αργότερα τον Επίτροπο Ιωάννης Χάν. Δεύτερο σημείο. Ανακοινώσει του Προέδρου. Αποφάσεις συντονιστών 12 Δεκεμβρίου. Είναι στο φάκελό σας αν θεωρούνται εγκεκριμένα. Καλώς. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων. Αν αντιδράσεων και αντιρρήσεων θεωρούνται εγκεκριμένα. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Ας ανασκουμποθούμε. Να δούμε τόσες ψηφοφορίες αν δουλεύει το μηχάνημα. Έχετε τις κάρτες ψηφοφοριών. Να κάνουμε μια δοκιμή. Εντάξει, άρχεται η δοκιμή ψηφοφορίας. Κυρία Χολμάιερ, εξακολουθούμε να έχουμε ανοιχτή τη διαδικασία. Μην βιάζεστε. Περιμένουμε. Πέρας. Ωραία, καλά τα πήγαμε. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε πρώτα απ' όλα μεταφορές τμήμα 3, ο κ. Χάουαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεταφορές του τέλους του έτους. Προϋπολογισμός 2019. Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται σε υποχρέωση πληρωμών Γίνονται αυτά για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα και να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Τα μεγαλύτερα στοιχεία ενισχύουν τρεις τομείς του προπολογισμού. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εδαφική Συνοχή φυσική πόρη, βιώσιμη ανάπτυξη, τίτλος 1, Γεωργία, Γεωργικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Μέσο για την Αλία και θαλάσσιες μεταφορές. Αυτές οι ανάγκες μεταφόρων, οι ενισχύσεις οικονομικές, οφείλονται στο ότι η κοινωνική και εδαφική συνοχή λειτουργούν πλήρως. Λειτουργούν πλήρως έχουν ρυθμό πορείας όπως το λέμε. Και καταφθάνουν οι λογαριασμοί για τα ταμεία. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει τον προπολογισμό φέτος προσεκτικά, ούτως ώστε οι πληρωμές να διατεθούν σωστά για το 2020. Εδώ μιλάμε βέβαια για τις περιόδους του 2019, παρομοίως. Γεωργία. Εκεί μικροπεσορμογές έχουμε πλευράς ποσοστίας. Βέβαια είναι μεγάλα τα κονδύλια για το Ταμείο Αλίας. Είναι ένα ταμείο που ανακτά τους κανονικούς ρυθμούς και αυτό το αντικατοπτρίζει η προσαρμογή. Καλό θα ήταν να παρακολουθούμε στο μέλλον τις εξελίξεις αυτές εξής πληρωμών αντισταθμίζονται από μειώσεις σε, άλλους, σε άλλες κατηγορίες του προπολογισμού. Διάφορα ποσά σε περιοχές όπου ήταν πιο αργή η εφαρμογή μέτρων από ό,τι αναμενόταν ή εκεί όπου η υλοποίηση ήταν κάτω σε εκτιμήσεις. Αυτό αφορά 33 γραμμές του προπολογισμού. Οι συνολικές αυξήσεις και ενισχύσει αφορούν 255,5 εκατομμύρια ευρώ και αντισταθμίζονται από αντίστοιχες περικοπές σε άλλε γραμμέ και εγώ συστήνω να υποστηρίξουμε αυτέ τι μεταφορέ. Ευχαριστώ κύριε Χάουαρντ. Κάποιο κοιόδη εισηγητή επιθυμεί να μιλήσει. Κύριε Σουρέο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχόλιων. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση με 21 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους εναντίον και 3 αποχές. Δράτω με τις ευκαιρίες να αποκλίνω κάπως από το επίσημό μας πρόγραμμα. Απευθύνομαι στον κύριο Χάουαρντ και τα τρία άλλα μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Συνεργάστηκα πιο στενά με τον κύριο Χάουαρντ οι τρεις Κυριακοί σίγουρα θα με συγχωρέσουν αν απευθυνθώ συγκεκριμένα στον κύριο Χάουαρντ. Κύριε Χάουαρντ, είναι η τελευταία σας παρουσία. Εδώ, δυστυχώς μπόρεσα να συνεργαστώ με τον κύριο Χάουαρντ μόνο για λίγους μήνες. Αλλά σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα διαπίστωσα ότι είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Χάουαρντ. Υπήρξε άνθρωπος πολύ ανοιχτός άμεσος με άριστη γνώση του αντικειμένου του και ευρύτερε γνώσεις από το αντικείμενό του βέβαια. Εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι ομιλώ εν ονόματι όλων ευχόμεθα σε εσά και στα άλλα τρία μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Επιτροπής Υπολογισμών, ό,τι καλύτερο. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε ότι τα δέντρα δεν συγκρούονται, αλλά οι άνθρωποι συναντώνται Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε κάποτε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Unfortunately, back to business. Um, Δυστυχώς τα τετριμένα τώρα. Ψηφοφορία δεν ζητήθηκε μεταφορά στο, στην κατηγορία 3 και στα άλλα τμήματα. Μπορούμε να πάμε στα κτίρια. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο κτίριο στο Πεκίνο. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο περί αυτού. Κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τρεις εκθέσεις έχουμε για τα κτίρια. Καταρχάς, ένα από τα κτίρια της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο. Υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εξετάσαμε εμπρότης το θέμα αυτό το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Θέλουμε να ανανεώσουμε τη σύμβαση. Για το North Wing, το κτίριο North Wing, έχουμε δύο κτίρια στο Πεκίνο, δύο τοποθεσίε, το North Wing για τέσσερα χρόνια. Ε, εν αναμονή ε, μιας οικοδομής στο South Wing. Υπάρχει και κτίριο, αλλά πολύ μικρότερο. Αλλά έχουμε ε, περιθώρια, οικόπεδο και σε 4-5 χρόνια μπορούμε να ενώσουμε όλες τις υπηρεσίες μαζί στην κτίριο. Το κτίριο για το οποίο ζητάμε την άδεια ανανεώσεως της μίσθωσης στεγάζει 75 άτομα, 50 της υπηρετησίας εξωτερικής δράσης, 8 μαθητευόμενους, 8 άτομα από άλλες ευρωπαϊκές δομές, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας Εναερίων Μεταφορών και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα πνευματικά δικαιώματα. Η έκθεση εμπεριέχει στοιχεία όσον αφορά το, το μίστομα. Έχουμε στοιχεία και αναφορές όσον αφορά την τιμή. Αυξάνεται η τιμή. Η αγορά στο Πεκίνο είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι σημαντικό να έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τα τι γίνεται με τις τιμές γύρω-γύρω. Τα τέσσερα χρόνια ε, ακολουθούν σχεδιασμό ρεαλιστικό. Για την οικοδόμηση του νέου κτηρίου, κατά 20% αυξάνεται το μίστομα και θεωρείται κάτι λογικό αν λάβουμε υπόψη της εξελίξεις στην αγορά. Ο συνάδελφος που γνωρίζει άριστα το θέμα, η κυρία Μόνικα Ολμάιερ, έθεσε πολλές ερωτήσεις και έχει μια ανησυχία ότι θα πρέπει να υποδεχθεί σε αυτή το εκτίριο υπηρεσία εξωτερικής δράσης και άλλου, Θα πρέπει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως να στεγαστεί ή να εκμεταλλευτεί αυτό το κτίριο τη υπηρεσία εξωτερική δράσης. Να υπάρξει συνεργασία. Πώς να το πω. Θα μπορούσε να υπάρχει βελτίωση στη σχέση μεταξύ διαφορών φορέων της Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Εγώ προτείνω να δεχτούμε αυτή την πρόταση, αλλά να το θέσουμε σημείο συζήτηση με την υπηρεσία εξωτερική δράσεω για να ληφθούν υπόψη όλε οι ανάγκε. Αποστολή μα να έχουμε καλή δημοσιονομική διαχείριση. Εκτό Βρυξελών και Στασβούργου να έχουμε μια ομαδική αντιμετώπιση όσον αφορά τι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή είναι πολύ καλό για του πολίτε. Προτείνω μια συζήτηση γενική προ αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πνεύμα, με την υπηρεσία εξωτερική δράσεω, τώρα στην αρχή τη θητεία, δείχνουμε θετική θέληση, καλή διάθεση προ όλου. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Κέλλερ. Κυρία Ολμάια. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Κέλλερ, σε μεγάλο βάθμο συμμερίζομαι την άποψη της συναδέλφου Κέλλερ. Έχω μια επίγουσα ερώτηση καταρχάς και εν συνεχεία να πω ότι αφού το συζητήσαμε μεταξύ μας υπάρχει ανάγκη να εγκρίνουμε, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια προϋπόθεση, δηλαδή να λυθούν ε, και να διευκανθούν κάποια ζητήματα μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Η ερώτησή μου καταρχάς είναι το πιο ακριβό ε, κτίριο ε, και με μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλο. και θα ανεβεί ακόμη η τιμή, η τιμή. Μετά έχουμε τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. και έχετε κάποια ποσοστά, 165, 140, Αυστρία, Ιρλανδία, ε, πάνω από 200 τόσα είναι στην ε, περίπτωση αυτή ε, η τιμή του κτηρίου σε σχέση με το τι πληρώνουμε που είναι κάτω από τα 200 στα άλλα ε, κράτη-μέλη το κτίριο. Δηλαδή 20% παραπάνω, ίσως και 30% παραπάνω από τα άλλα κτίρια των άλλων πρεσβειών στο ίδιο ουσιαστικά επίσης μέρος γη στην ίδια περιοχή. Αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά την ε, ΕΙΕΔ και το Κοινοβούλιο ότι ίσως δεν έφερθήκαμε, λένε πάρα πολύ φιλικά και τους έχουμε θέσει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Ε, ε, έχουμε το κτίριο στο Λονδίνο. Αρχικά για αυτή η προσπάθεια να το πάρει από το κοινοβούλιο αυτό το κτίριο, να στερηθούμε ουσιαστικά δηλαδή ένα δικό μας περιουσιακό στοιχείο, αλλά ήταν δικό μας αυτό το περιουσιακό στοιχείο και δεν θέλαμε να το χάσουμε. Εκεί υπήρξε συνεννόηση. Το δεύτερο είναι ότι η ΕΕΔ, η εξωτερική υπηρεσία, θέλουν να έχουν αποσπασμένους εθνικούς υπαλλήλους. Και αυτό έχει να κάνει με συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου από τον Ιούλιο του 2010 για μια συμφωνία συνεργασίας αντίστοιχη με αυτή που έχουμε στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή να είμαστε στο ίδιο κτίριο με την και σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι αποσπασμένοι εθνικοί υπάλληλοι από τα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά ε, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. εμείς ως Κοινοβούλιο ε, υποτίθεται ότι είμαστε ε, αρμόδιοι να πληρώνουμε ε, τους υπαλλήλους ε, σε ένα τρίτο κράτος. Υπάρχει επίσης απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Αφρικανική Ένωση και την ΑΣΕΑΝ να υπάρχει ε, αυτή η προσπάθεια για μια ευρύτερη συνεργασία Γι' αυτό είχαμε πάρει αυτή την απόφαση και για τη στέγαση των υπηρεσιών ε, της ΕΕΔ στις πρεσβείες. Αλλά ε, δεν θέλουμε να δούμε τι γίνεται... Ε, μάλλον δεν θέλουμε να πετούνται περισσότερα κονδύλια από εμάς ε, ξέρετε τι γίνεται και με την ΕΤΕΠ, για παράδειγμα. Εγώ ε, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, υπάρχει ναι, και οι γραπτές αποφάσεις και οι γραπτές συμφωνίες. διότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την υπογραφή, να λυθεί το πρόβλημα και να δώσουμε την έγκρισή μας για το Πεκίνο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τόσο φιλικοί γιατί θα είναι σε βάρος μας. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Πρέπει να βάλουμε ε, αυτές τις τέσσερις προϋποθέσεις. σε σχέση με Ασιαν Λονδίνο, Αφρικανική Ένωση. Ε, αν έχουμε τις τέσσερις προϋποθέσεις οποίες γράφω και συμφωνήσουν, τότε μπορούμε να εγκρίνουμε και το Πεκίνο. πράγματι υπήρξε ίσως όχι τόσο φιλική συμπεριφορά, αλλά τα διπλωματική και πάντα μέσα στα όρια. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε και τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα ως κοινοβούλιο και όχι να υποχωρούμε απέναντι στην τώρα θα ήταν λιδία λίθος αν θέλετε η περίπτωση του Πεκίνου για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε να υιοθετηθούν αυτές, αυτά τα αιτήματά μας οπότε να εγκρίνουμε και το Πεκίνο. Εγώ έχω δει ε, και τις συμφωνίες, ε, έχω δει τις συνθήκες. Ε, υπάρχουν ουσιαστικά υπογραφή λύπη και εμείς νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στην εκπλήρωση αυτών των τεσσάρων ε, όρων και προϋποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια. Στεφανούτα. I only wish to take the floor. Όχι, θέλω το λόγο ε, για να πω απλά ότι ε, εμπιστεύομαι τις ε, κυρίες Κέλλερ και Ουάσιγκτον στην προηγούμενη θητεία είχε πει το Κοινοβούλιο ότι θέλει να εκπροσωπείται σε τέσσερα μέρη του κόσμου, την Ουάσιγκτον, εκεί έχουμε γραφείο, κοινό με την ΕΕΔ και έχουμε καλή συνεργασία. Το δεύτερο θα ήταν ε, στην Αντισαμπέμπα, το τρίτο στην Τζακάρτα για την Ανατολική Ασία και το τέταρτο νομίζω είναι για την ΟΙΕ στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε προσπάθησε ε, συνεχώς η ΕΕ να μπλοκάρει τις εξελίξεις, δεν δίνει έγκαιρα ε, για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν εκεί και γι' αυτό θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι καλή διοργανική συνεργασία και μπορεί να παίξει καλύτερο ρόλο. Πιστεύω το Κοινοβούλιο σίγουρα είναι πολύ στενά τα νοσονομικά όρια που έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να μας ε, φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρος, άλλα σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε σιγά σιγά. Anybody else? We have uh, Madame Vasquez Garrido of... Είναι κάποιος από την ΕΕΔ εδώ και Έχουν τεθεί πολύ σοβαρά ερωτήματα και ζητήματα. Θα ήθελα η εκπρόσωπος της ΕΙΔΕ που είναι εδώ να μας πει αν μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Δεν έχω πολύ το τίποτα να προσθέσω σε αυτή την παρουσίαση της εισηγήτριας, της κυρίας Κέλλερ. Κάμια πολύ καλή σύνθεση της υπόθεσης, άρα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα της κυρίας Χολμάιερ, δεν είναι τόσο μέσα στο δικό μου πεδίο αρμοδιοτήτων. για το κατά πόσο, μάλλον γιατί είναι τόσο ακριβό το κτίριο αυτό, σε σχέση με αυτό το ερώτημα, γιατί είναι το πιο ακριβό ανά ε, τετραγωνικό μέτρο. Δεν ξέρω. Τα στοιχεία που έχουμε δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι το πιο δαπανηρό κτίριο. Έχω εδώ κάποια στοιχεία για να σας πω περίπου τι πληρώνουμε σε άλλε περιπτώσει. να μπορεί να μου πει ποιο είναι ο μεσοσόρο. παρακαλώ. Θα έλεγα ότι είναι και κάτω από το μέσο όρο. Ναι, είναι κάτω από το μέσο όρο. Ο μέσο όρο. είναι 3,53 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και για το δίκτυο είναι 435. Άρα κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ υπήρξε ίσως κάποια παρανόηση. Και η πιο ακριβή αντιπροσωπεία είναι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα δεν είναι αυτά τα στοιχεία ακριβή. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν άλλες πρεσβείες που πληρώνουν χαμηλότερες τιμές στην ίδια περιοχή. Αυτό εξαρτάται από το πότε συνάφθηκε η μίσθωση. Γιατί είναι η αγορά των ακινήτων πάρα πολύ ρευστή και τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Ολόκληρες γειτονιές. Ε, πριν να κλείσει τα μάτια σου, ε, έχουν αντικατασταθεί τα κτίρια εκεί από σύγχρονα και έχουν ανέβει τιμές. Επομένως, ανάλογα με το πού και πότε ε, έχει υπογράψει κάποιος ε, τη σύμβαση της μίσθωσης, μπορεί να αλλάξει εντελώς η τιμή. Εμείς σίγουρα προσπαθούμε να ελέγχουμε τις τιμές τη αγοράς για να έχουμε κάποιε συγκρίσιμε τιμέ. Δεν έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία για την ποιότητα των άλλων ε, κτίριων. Τώρα, αν είναι πιο χαμηλής ποιότητα από αυτά τα οποία μισθώνουμε εμείς, φυσικά και θα είναι και ε, πιο φθηνά. Πάντως, κάναμε αυτή την ανάλυση και η τιμή νομίζω είναι συγκρίσιμη με τη μέση τιμή των κτίριων ε, της ίδιας ποιότητας. Τα άλλα όμως ερωτήματα δεν είναι της δικής μου ευθύνης και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για αυτά. Ο Χέλγα Σμιτ, Γενική μας Διευθυντήρια και Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου, τα συζητούν αυτά. Δεν θα επισέλθω σε σχόλια για μια συζήτηση που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Πάντως θέλουμε να υπάρξει ε, ξεκαθάρισμα οποιονδήποτε παρανοήσεων και κάναμε μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες. Παρά τη μεγάλη περίοδο σιγής επικράτησε δυστυχώς για μεγάλο διάστημα μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Αλλά η σχέση βελτιώνεται και μάλιστα τάχιστα. Και έτσι πολλές από τις παρανοήσεις που υπήρχαν έχουν διασκεδαστεί, ότι δηλαδή η ΕΕ ζήτησε να πεμπολίσει σε κάτι στοιχεία το Κοινοβούλιο. Όχι βέβαια σε καμία περίπτωση. Αυτό ήταν παρανόηση και νομίζω έχει διευκρινιστεί και θα βρεθεί λύση το είπε και η Τώρα δεν έχω εξοδότηση για να μπω σε συζήτηση ό,τι αφορά προσωπικό, τους υπαλλήλου. Είμαστε όμως υπεύθυνοι για την ε, συγκατοίκηση εντό αγωγικών, όπως με την ΕΤΕΠ, την ε, τράπεζα που αναφέρθηκε ως παράδειγμα. Και εδώ όμως έχουμε μια παρανόηση. Πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΕΠ δεν εντάσσεται στις αντιπροσωπείες έχουν ανεξάρτητη παρουσία στις τρίτες χώρες. Αυτό προβλέπεται από το καταστατικό και ανάλογα με τις διευθετήσεις που έχει η χώρα έχουν δικές τους συμφωνίες με βάση τη σύμβαση της Βιέννης. Είναι ανεξάρτητη η παρουσία τους εκεί. Ανεξάρτητη και από ε, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντιπροσωπείες. και από την ΕΕ που εγώ. Το μόνο που γίνεται είναι ότι διευκολύνουμε την παρουσία τους στο κτίριο, στις εγκαταστάσεις, χωρίς να τους προσφέρουμε καλύτερους όρους όμως. Εφαρμόζουμε τα εισήριας ε, ακριβώ ε, τιμές. Είναι ουσιαστικά διοικητική η μόνη διευθέτηση. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, αυτές όλες οι συζητήσεις που γίνονται, ε, που είναι πολιτικές όμως και εγώ δεν μπορώ να τις σχολιάσω. Αλλά σίγουρα δεν επιφυλάσσουμε χειρότερη μεταχείριση ε, στο κοινοβούλιο οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό εταίρο. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ότι θέλετε να με ρωτήσετε για αυτό το project, για την αντιπροσωπεία στην Κίνα. Thank you. Does uh, anybody... Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Το κείμενο το οποίο σας προτείνει η κυρία Χολμάιερ ε, τη ζήτησαν το διανύμι και σε όλες οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Και βέβαια δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από τους αντιπροσώπους Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να το εγκρίνουν εδώ και τώρα. Πάντως, αν συμφωνείτε με το κείμενο αυτό, μπορεί να πάρει το λόγο κυρία Χολμάιρ πρώτη και έπειτα η συγκίτρια κυρία Κέλλερ. Για τις τιμές καταρχάς. Προσπαθείτε να τα πείτε διπλωματικά και φυσικά και είναι το ισχυρό σας σημείο ως ε, αλλά δεν μιλάμε για ε, κάποια κτίρια έτσι χαμηλότερης ποιότητας ή αξίας. Πρόκειται για πρεσβείες. Ε, είναι στο ίδιο μέρος, στην ίδια περιοχή και δεν πρόκειται για φθηνότερα, λιγότερο ποιοτικά κτίρια. Ταλία, Βέλγιο, σας είπα, Πορτογαλία επίσης, Αυστρία ε, δεν ε, είναι τίποτα τρόγλες και μαζί με όλους τους συναδέλφους θα ε, ήθελα και εγώ ως το συντομότερα να εγκρίνουμε το Πεκίνο. Αλλά έχουμε συνέχεια αυτό το θέμα με τα τετραγωνικά. Εδώ και 11 χρόνια το συζητάμε. Υπάρχουν όμως και άλλες πρεσβείες ή αντιπροσωπείες ε, που στην ίδια περιοχή ε, έχουν κτίρια με πολύ χαμηλότερες τιμές έχουν το table of office premises of member states indicating in particular the size and the rent. Ότι αναφέρεται το μέγεθος, αναφέρεται η τιμή. Άρα ξέρω που είναι, τι τιμή έχουν οι πρεσβείες, γι' αυτό και η απάντησή σας ε, δεν με ικανοποίησε για να πω την αλήθεια μου. Το δεύτερο. Θα ήθελα προς όφελος όλων των συναδέλφων και εισηγητών. Να πω ότι ήδη από τον Ιούνιο ε, έχετε όλες τις διευκολύνσεις και το πήραμε και εμείς αυτό το φάκελο πρόσφατα θα ήταν καλό να είχαμε χρόνο για να μελετήσουμε όλα αυτά τα έγγραφα και όχι η ΕΕΔ να μας λέει ότι υπάρχουν τώρα αυτά τα ε, έγγραφα, αυτός ο φάκελος. Πράγματι, τα είχαμε από τον Ιούνιο, υποτίθεται αυτά τα έγγραφα, αλλά καλούμαστε να πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα αποφάσεις και αυτό δεν προωθεί την ε, εμπιστοσύνη. Ούτε είναι καλό να μας λέτε ότι αν το Πεκίνο δεν εγκριθεί θα είναι πολύ άσχημο και θα φέρετε την ευθύνη ως κοινοβούλιο. Όχι, συγγνώμη. Ε, για το κείμενο το δικό μου ε, που ε, νόμιζα ότι το είχατε όλοι, ε, δεν το ήξερα ότι δεν τα έχετε πάρει αυτά τα τέσσερα σημεία για τα οποία μιλούσα. Βεβαίως και θα το ε, διαβιβάσω ε, σε όλους τους συναδέλφους, αλλά συνάδελφος από τη Ρουμανία που δεν ξέρω πώς λέγεται. Στέφανου, πώς λέγεστε. Τέλος πάντων, καλά, θα το βρω. Στεφανούτα, κάπως έτσι. Ναι, ε, για να μην το πω λάθος το όνομά σας. Και με τον κύριο Πέξα ε, τον ε, αλλά υπάρχει και μία λέξη έτσι όχι και τόσο ευγενική ε, στα τσέχικα που προφέρεται ακριβώς έτσι, λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, αν επαναλαμβάνω αυτά τα τέσσερα σημεία γίνουν αποδεκτά, τότε μπορούμε να εγκρίνουμε αυτομάτως και το Πεκίνο. Η κυρία Κελέρα. Θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω επίση και του συναδέλφου και όλου ιδιαίτερω την Μόνικα που γνωρίζει πολύ καλά το φάκελο αυτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν για τι παρατηρήσει σα και για το ότι παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυ την υπόθεση αυτή. Να ευχαριστήσω βέβαια και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τα στοιχεία που μα έδωσε. Κάποια συμπληρωματικά στοιχεία από μένα τώρα πρέπει να επιβεβαιώσω και προς την ΕΙΕΔ ότι υπάρχει όντως ένας πίνακας όπου έχουμε τις διαφορετικές πρεσβείες και την τιμή είναι τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για πρεσβείες οι οποίες από ό,τι φαίνεται καταβάλουν μια τιμή χαμηλότερη από αυτή που μας προτείνεται. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Είμαστε όμως στην Κίνα και θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσο θα διαρκήσουν οι μισθώσεις αυτές, ποια είναι η φύση των κτηρίων αυτών. Ξέρετε όπω και στην Ελβετία Πρόκειται για μισθώσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα μακροχρόνιες και δεν ακολουθούν εδώ πέρα οι τιμές ακριβώς τους κανόνες όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ πέρα έχουμε μισθώσεις βραχίε, βραχίες, τεσσάρων ετών. Έχουμε πάντως και ένα κείμενο, ένα έγγραφο μάλιστα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, το οποίο περιγράφει την το διαγωνισμό που έλαβε χώρα προκειμένου να αποκτήσουν το κείμενο αυτό. 13 προτάσεις έλαβαν, εκ των οποίων 5 τις ανέλησαν ακόμα περισσότερο γιατί ανταποκρίνονταν περισσότερο στην προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το έγγραφο λοιπόν αυτό είναι πιο πλήρες και ανταποκρίνεται λίγο περισσότερο στην προτινόμενη τιμή. Ενδεχομένως λοιπόν ανταποκρίνεται λίγο περισσότερο στην πραγματική εικόνα τη ε, στεγαστική αγορά όσο έχει αυτή τη στιγμή στην Κίνα, βάσει τη φύση του κτηρίου και τη διάρκεια τη μίσθωση που επιθυμούμε. Και το είπα άλλωστε αυτό και εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ότι η στεγαστική αγορά παρουσιάζει τεράστιε διακυμάνσει, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη. Δεν ε, μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να ξεκινούμε πάντα τη διαδικασία από το μηδέν. Θα πρέπει να βρούμε μια πιο ρεαλιστική, πραγματιστική λύση και εν να καταφέρουμε εμεί τώρα να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα γραφεία του Πεκίνου. Βέβαια, κρεμεί το ζήτημα του Λονδίνου, διακόπτει ο πρόεδρο. Πρέπει να ψηφίσουμε όμω κάποια στιγμή, κυρία Κέλλερ. Θα αναλύσουμε λίγο αργότερα το Λονδίνο, αλλά πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε για το Πεκίνο. Προτιμάτε μετά, κύριε Πρόεδρε. Ναι, προτιμώ. Απλώς ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση της κυρίας Χολμάιερ και στο εγγραφό της. Για το Λονδίνο πάντως θα εμβαθύνω λίγο περισσότερο στο ζήτημα αυτό και εν ευθέτω χρόνο θα σας κάνω και μία παρουσίαση. Όσον με αφορά πάντως απευθύνομαι και στη Μόνικα, τώρα μόλις ξεκινώ να ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό, εσείς το γνωρίζετε πολύ περισσότερο. Έχουμε ένα νέο εκπρόσωπο, ένα νέο επικεφαλή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Με αυτόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μία ει βάθο συζήτηση όσον αφορά την μέθοδο που θα ακολουθηθεί στο μέλλον. Όντω, τα έγγραφα μα δόθηκαν τελευταία στιγμή. Δεν ελήφθη υπόψη η έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορεί να εκπροσωπείται περισσότερο στην όλη αυτή τη διαδικασία και σε συγκεκριμένε 5-6 τοποθεσίε στον κόσμο. Η κυρία Χολμάιρε πάντω έκανε μια πολύ καλή εργασία και νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε το εγγραφό της, να λάβουμε γνώση των πληροφοριών που μας δίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει το έγγραφο αυτό να αποτελήσει μια καλή βάση για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και συνεργασίες που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ζητώ μόνο να μου δώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να μπορέσω στο μέλλον να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κτηρίων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάρα έχει το λόγο. Δεν είναι επιλογή αυτή για μένα. Είχαμε αποφασίσει ε, όταν συνομιλήσαμε κατηδίαν μαζί, κυρία Κέλλερ, ότι θέλουμε σήμερα να ψηφίσουμε ουσιαστικά να πάρουμε την απόφαση και με βάση αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν έχουμε νομίζω πλέον ε, βάση. Με αυτή τη συζήτηση δηλαδή που έγινε σήμερα με την ΕΙΕΔΕ δεν έχουμε κάποια βάση. Ε, νομίζω ότι ως κοινοβούλιο πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούν ε, να μας ε, φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε σε μία συμφωνία Εμείς είμαστε ε, φιλικοί, αλλά ουσιαστικά δίνουμε ε, όχι τις τιμές της αντικειμενικές της αγοράς, αλλά κατά κάποιο τρόπο ιστορικές τιμές. Ε, αυτές είναι οι τιμές των συμβάσεων, συμβάσεων μίσθωσης, τελείως διαφορετικές τιμές στο Λονδίνο σήμερα ε, τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει προσωπικό το οποίο θα θεωρείται αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Ε, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να το δεχθούμε. δεν μπορεί να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκπροσωπείται σε άλλες χώρες. Ε, όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Προσπαθούμε επί μήνες ε, να βρούμε μια λύση ε, και νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε και πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά τα σημεία για να υπάρξει κάποια αντίδραση, να υπάρξει κάποια επιτάχυνση της διαδικασίας διότι στην Ουάσιγκτον έχουμε αυτή τη συγκατοίκηση εντό αγωγικών. Τα είπε ο συνάδελφο από τη Ρουμανία πάρα πολύ καλά ε, και λειτουργεί και βασίζεται και στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και τώρα η ΕΕΔ προσπαθεί ουσιαστικά να μα ε, ε, κάνει να γυρίσουμε πίσω σε μια άλλη κατάσταση. Όχι. Συγγνώμη που τα λέω τώρα έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Σας παρακαλώ να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε έτοιμες αυτές τις συμβάσεις, μπορούμε να τις υπογράψουμε όποτε θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν να ασκούνται πιέσεις στο Κοινοβούλιο. δεν θα ήθελα να εγκρίνουμε το Πεκίνο έτσι χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση γιατί αυτό θα δείξει αδυναμία απέναντι στην ΕΕΔ. Τέλο πάντων, ε, με βάση ε, το, τι γίνεται στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε αντίστοιχα να αποφασιστεί για την Τζακάρτα, την Αντισαμπέμπα και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Την ίδια βάση θέλω ότι ισχύει για την Ουάσιγκτον. Εγώ δεν θέλω κάτι διαφορετικό. Ε, η δεν θέλει να μας τριμώξει σε μια χειρότερη θέση. Εγώ θέλω την ίδια θέση. Και υπάρχει αυτή η απόφαση του 10 από το Συμβούλιο, την οποία την έχει δεχτεί και η ΕΔ. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει δοθεί κατάλληλη απάντηση στα ερωτήματα που ετέθησαν. Εξίσου σαφές είναι ότι σε διάφορα επίπεδα υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας, όμως ε, πρέπει να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εγώ τι προτείνω. Να κάνουμε δύο ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα για το Πεκίνο, τελεία και παύλα. Και δεύτερον, αν τα τέσσερα σημεία, όπως τα παρουσίασε η κυρία Χολμάιερ, αν τα θεωρούμε ότι εξαρτώνται από την πρώτη ψηφοφορία. Πρώτα το Πεκίνο και μετά το άλλο. Η κυρία Κέλλερ. Διαρωτώ με αν πρέπει να ψηφίσουμε στο δεύτερο σημείο. Δεν λάβαμε γνώση του εγγράφου, δεν μεταφράστηκε κλπ. Με μια ματιά βλέπω ότι θεωρούμε ότι συμφωνούμε. Πρώτη παράγραφος είναι έχουμε παρουσία στο Λονδίνο. Δεύτερο, στη δεύτερη υπενθυμίζει αυτός που έλεγε ο συνάδελφος Στεφανούτα, παρουσία στην Τζακάρτα, Αντίσα Μπέμπα, Ουάσιγκτον. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τέταρτη υπενθυμίζουμε την κατάσταση στο Λονδίνο, αναφέρονται διάφορες αρχές και ότι στα τέσσερα γραφεία του κόσμου πρέπει να είμαστε κατάλληλα δεκτοί. Πρέπει να προσθέσουμε και το Λονδίνο. Έχουμε τέσσερι τοποθεσίε, αλλά πέντε. Θα έλεγε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ότι δεν είναι πλέον εκεί. Καταρχήν, θεωρώ ότι το πακέτο έχει δυσκολίες θα μ' άρεσε να μπορούσαμε να ψηφίσουμε επί ενός κειμένου το οποίο το έχουμε επεξεργαστεί κάπως, το έχουμε κουβεντιάσει. Δεν είχαμε το έγγραφο. Θα ήταν κρίμα να ψηφίσουμε. Όπως θέλετε κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αποτελεί βάση εργασίας. Μπορούμε να ψηφίσουμε ότι αποτελεί βάση εργασίας που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Πρόεδρος. συζήτηση με την υπηρεσία εξωτερική δράση. Τι λέτε, ότι οι συνθήκε δεν είναι όπω αυτέ. Ότι αυτέ όπω παρουσιάζεται το έγγραφο οι συνθήκε δεν θα έπρεπε να δημιουργούν πρόβλημα. Αντί αυτή η περίπτωση και το να εξαρτάται το δεύτερο σημείο από το πρώτο δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Να πω καταρχά. Στι 11.30 έχουμε τον κύριο Μάριτ και άλλα σημεία. Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε τώρα εσαΐ να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω την πρότασή Ψηφίζουμε το Πεκίνο και μετά τέσσερα σημεία, εξαρτώμενα από το ε, Πεκίνο. Madame Guardia Zabal. Sí, gracias, presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα παράλληλα μια άλλη συνεδρίαση και δεν παρακολούθησα τις συζητήσεις μέχρι τώρα, όμως... Ότι είχε συζητήσει η συγγήτρια με την ΤΕΟΣ, καλό, είναι εντάξει. Αλλά εμείς δεν είμαστε ενημερωμένοι για το έγγραφο, για τίποτα. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ε, να έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί τώρα, να, διαβάσουμε, να αναλύσουμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας αν η ομάδα μας συμφωνεί όχι, δεν επαρκεί ως χρόνος τώρα. Καλώς. Υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα. Ας το ξανακουβεντιάσουμε το απόγευμα, αφού έρθει ο κ. Χάν να ψηφίσουμε τώρα στις 11 ή στις 5 το απόγευμα δεν κάνει διαφορά. Μέχρι τότε όλοι θα έχετε το χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά τις 20 γραμμές. Μόνο 20 γραμμές είναι, δεν 20 σελίδες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα θα πρέπει κανονικά να είμαστε έτοιμοι να το εξετάσουμε το θέμα κανονικά όπως το αρμόζει και να λάβουν χώρα και συζητήσεις που δυστυχώς δεν έλαβαν χώρα νωρίτερα. Ψηφίζουμε το απόγευμα για το Πεκίνο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κτηριακή πολιτική και ανταλλαγή απόψεων. Πάλμερστον. Το κτίριο Πάλμερστον εδώ στις Βρυξέλλες. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι, ε, το Frontex είναι, είναι βρεθικό σταθμός, τι. Πάλμερστον. Τα, μαζί, λέει ο πρόεδρος, να τα πούμε είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε σαν βρεφικός σταθμός και έγινε επίσης και νηπιακό σταθμός για μετά το σχολείο. Κάποια ενημέρωση αρχική είναι αυτή. Προτείνεται ανοικοδόμηση βρεφικού σταθμού μεταξύ από διάφορε χρήσει του κτηρίου που δεν είναι πλέον σε πολύ καλή κατάσταση, χρειάζεται ανακαίνιση σημαντική. Για να μπορεί να δέχεται τα μικρά παιδιά δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για την ώρα. Είναι πολύ διαφορετικό το θέμα από το θέμα Frontex. Απλώς έγκαιρη προειδοποίηση είναι αυτή. Ήδη είναι καλή βάση για να την επεξεργαστούμε ήρεμα για τελική παρουσίαση. Το κτίριο θα μπορεί να δέχεται παιδιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σύμφωνα με τους κανόνες για τη μέρη με των παιδιών του προσωπικού προτείνω θετική αντιμετώπιση. Καλό θα ήταν να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτού του είδου τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Βλέποντα το χρόνο που μας απομένει, δεν θα συζητήσουμε πλήρως το θέμα. Τώρα θα επανέλθουμε αργότερα όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. κυρία Κέλλερ για τη Βαρσοβία, την κεντρική μας μονάδα εκεί. Ναι, πράγματι, Πρόκειται για την οικοδομή, για να βρούμε μια νέα υποδομή για το αιτίας, την υπηρεσία Το νέο σύστημα πληροφοριών που θα έχει τα στοιχεία, τα δεδομένα, το αιτίας, για τη διαχείριση των θεωρήσεων και επιχειρησιακή λειτουργία των δεδομένων. Το κτίριο αυτό έχει κάποια στοιχεία πληροφορικής, κάποιο εξοπλισμό πληροφορικής και προσωπικό. 24 ώρες το 24ωρο θα εργάζεται. Σε πραγματικό χρόνο θα υπάρχει διαβούλευση με τη βάση δεδομένων για τη διέλευση συνόρων. Και θα εγκατασταθεί όχι πολύ μακριά από την έδρα της Frontex στη Βαρσοβία στενή συνεργασία υπάρχει με άλλου χειριστέ. Το EU LISA που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Υπάρχει διαλειτουργικότητα, διασύνδεση μεταξύ αυτών των συστημάτων και των βάσεων δεδομένων. Απλώ ναι, για λάβετε γνώση, αρχικέ πληροφορίε. Δεν θα είναι το τελευταίο θέμα η τη Frontex. Θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητε περαιτέρω τα επόμενα χρόνια τη Frontex. Ήδη προβλέπεται για τον προπολογισμό του 2020, όχι πάντα στη Βαρσοβία αλλά και στα κράτη-μέλη για να, είναι, να υπάρχει εγκύτητα του προσωπικού με τις χώρες, η Frontex μας παρουσίασε μια στρατηγική 2019-2024 Πολύ πρόσφατα έθανε οι πληροφορίες, δεν τις έχω εξετάσει διεξοδικά. Μπορώ να τις διαβάσω στα μέλη. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά όσον αφορά το σχεδιασμό και την βελτίωση της ισχύω του όλου μηχανισμού Frontex και όλων των συναφών δομών, όπως το αιτίας εδώ. Θετική γνωμοδότηση και μπορούμε να το εξετάσουμε αρκετά ε, γρήγορα και σύντομα. Είναι το κτίριο για το αιτίας λοιπόν. Ευχαριστώ. Τα ίδια σχόλια λοιπόν, όπως και για το Palmerston. Θα επανέλθουμε αργότερα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Στονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, ε, τη επισκόπηση τη ανάπτυξη για το 2020. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρκη για να μα παρουσιάσει εν συντομία το σχέδιο γνωμοδότησή τη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέσατε πολύ σωστά. όντω η παρουσίασή μου θα είναι πολύ σύντομη. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση και καθότι πρόκειται για γνωμοδότηση αποφάσισα να έχω μια προσέγγιση μινιμαλιστική. Και προφανώς μπορείτε μέχρι τις 28 Ιανουαρίου να καταθέσετε όσο το επιθυμείτε τροπολογίες. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν έχω συμπεριλάβει 7 σημεία. Πρόκειται για κάποιες προτάσεις τι οποίε θα θέλαμε να λάβει υπόψη στην τελική τη έκθεση η Επιτροπή οικονομική και Νομισματικής πολιτική ΕΚΟΝ. Στο πρώτο σημείο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη για να ανταποκριθεί στις περιβαλλοντικέ κλιματικέ, ψηφιακέ και δημογραφικέ προκλήσει. Και λέμε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει σε μία πράσινη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ευρώπη. Δεύτερη πρόταση. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι όλες αυτές οι προκλήσεις θα έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις κοινωνίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όταν αφαιρόμαστε στα κοινωνικά δικαιώματα και στις ανισότητες. Γι' αυτό λοιπόν, ακριβώς το λόγο, στο δεύτερο σημείο της γνωμοδότησής μου, προτείνω, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να εφαρμόσουμε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. και στο ίδιο πλαίσιο, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες ανησυχίες, λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης στις αναχώρα εκθέσεις. Στις αναχώρα συστάσεις μάλλον. Τώρα, όσον αφορά τις εκθέσεις επιδόσεων της ενίας αγοράς, Νομίζω ότι οι εκθέσεις αυτές πραγματικά θα καταδείξουν τα ωφέλη της ενίας αγοράς για τα επιμέρους κράτη-μέλη και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο με τις εκθέσεις αυτές θα καταφέρουμε να καταρρύψουμε τους μύθους που υπάρχουν γύρω από την προσέγγιση των καθαρών συνεισφερόντων και των καθαρών αποδεκτών. Αναφερόμαστε επίση σε διάφορους στόχους, στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότερο στην κατάρτιση της μεθοδολογίας η οποία θα πλαισιώσει οποιαδήποτε δαπάνη κοινοτική θα γίνει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η μεθοδολογία αυτή βέβαια θα πρέπει να καταρτιστεί, θα πρέπει να θεσπιστεί, θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανής Και αν καταφέρουμε στα πλαίσια τη μεθολογία αυτή να έχουμε ποστικοποιημένου στόχου, θα πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη μεθολογία για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχου αυτούς. Άρα λέω για μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέξει στην όλη αυτή τη διαδικασία περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα στο έκτο σημείο τη γνωμοδότησή μου λέμε ότι ε, οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάνε από διαφορετικά σημεία κίνηση όσον αφορά τι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επομένω, ο περίφημο μηχανισμός δίκης μετάβαση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η μετάβαση αυτή θα είναι κατάλληλη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμού για όλες τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβδομο τέλο σημείο. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο τη δημοκρατική λογοδοσία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος από τους κοιόδης ηγητές να πάρει τώρα το λόγο. Ρέσλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την συντάκτρα της γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση αυτή και όλες τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα εργαλείο όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο θα προσφέρει μια διαφανή, ένα διαφανή συντονισμό πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διαφορετικές μεταρρυθμίσει που έχουν ως στόχο κυρίως την κοινοτομία, την έρευνα, την ψηφιοποίηση, τι επενδύσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και ένα βιώσιμο περιβάλλον. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο τελικά θα έχουμε μια πιο ανταγωνιστική και πιο πράσινη φιλοπεριβαλλοντική οικονομία. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε ισότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση χωρίς αποκλεισμού για όλες τις περιφέρειες, για όλες τις περιοχές και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει αυτό να φαίνεται και από την ίδια τη χρήση του κοινοτικού προπολογισμού. Τώρα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η οικονομική στρατηγική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων. Θεωρούμε επίση ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μοντέλα για να αντιμετωπίσουμε τις δημογραφικές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε τέτοια πρότυπα, τέτοια μοντέλα και θα πρέπει και αυτά να συμπεριληφθούν στο νέο βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Μετά, αγαπητοί συνάδελφοι, από αυτά που ακούστηκαν. Έχω κάποιες επιφυλάξεις, όχι σε ό,τι αφορά τις διαπιστώσεις για τα μακροοικονομικά αποτέλεσματα που είναι αρνητικά με χαμηλούς ποσοστούς ανάπτυξης, 1,4 του ΑΕΠ για το 19, ένα-δύο ο προπληθωρισμός για Γαλλία και άλλες ε, χώρες ε, πολύ χρέος, 90% στην περίπτωση της Γαλλίας και ένα στους πέντε Ευρωπαίους ε, ε, κάτω από το κατόφλι της Και αυτό πραγματικά μου φέρνει ρίγιο σε σκέψη. Έχουμε και την δημοσιονομική θέση για την Ευρωζώνη. Μια ιδέα που έχει ως στόχο να ευνοεί μεταφορές πιστώσεων για την αντιμετώπιση ασυμμετρών κραδασμών. Εγώ ως Ευρωβουλευτής οφείλω να προειδοποιήσω τους συμπατριώτες μου για το κίνδυνο να χάσει πολλά δις ευρώ η Γαλλία από αυτό. Υπάρχουν συνάλληλοι που μας εξηγούν για τους καθαρούς συνεισφέροντες που ωφελούνται από την αγορά. Όμως μόνο η Γερμανία είναι αυτή. Ουσιαστικά, στο πούμε ξεκάθαρα, στη Γαλλία και χάνουμε 8 δις ετησίως λόγω του ευρωπαϊκού προβλησμού, αλλά έχουμε και εμπορικό έλλειμμα ε, απέναντι στην Ένωση. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική και εφορική εναρμόνιση. Η Ένωση θέλει να δημιουργήσει πράγματα που δημιουργεί η ίδια όμως. Έχουμε χώρες στην Ενία αγορά ε, που διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους ε, και πώς μπορούμε να τα ισορροπήσουμε όλα αυτά. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να αρμονίσουμε τη φορολογία και να έχουμε ένα κατώτατο μισθό. Και εδώ έχω τις αμφιβολίες μου σε ό,τι τώρα αφορά τι συστάσει της Κομισιόν προ τα κράτη-μέλη, που είναι οδηγίε, εγώ θα έλεγα, πιο πολύ εντολές. Και πρέπει ε, ουσιαστικά να τις υποχρεώνουμε τις χώρες να τα εφαρμόζουν αυτά, αυτές τις εν λόγω συστάσεις. Και αλλιώς έχουμε τις ε, διαδικασίες ε, υπερβολικού ελλείμματος ή αναστολή χρηματοδότησης. Στη Γαλλία έχουμε τη μετα... μεταρρύθμιση του αξιοδοτικού συστήματος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπερεθνικός φορέας ε, που θα μπορούσε να μας υποκαταστήσει. Εμείς ξέρουμε καλύτερα και όχι αυτά που έχει αποφασίσει η Κομισιόν το 18-19. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τη συντάκτρια γνωμοδότη, την κυρία Μαρκέ, για την γνωμοδότησή τη αυτή με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ ότι όντω θα πρέπει να ακολουθήσει μια νέα πολιτική, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι η όλη δημοσιονομική διαδικασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τι συστάσει αυτέ τι οποίε προτείνει η κυρία Μαρκέ. Ισορροπημένη λοιπόν η προσέγγιση τη συντάκτρια γνωμοδότηση και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω το λέει, να μην μείνει κανεί εκτό διαδικασία αυτή. Άρα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και θα πρέπει επίσης να έχουμε έτσι έναν ισχυρό, αξιόπιστο, φιλόδοξο προϋπολογισμό, όπως άλλωστε έχουμε πει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και νέοι οι ίδιοι πόροι. Μόνο λοιπόν να ακολουθήσουμε τι παραμέτρου αυτή, θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την κλιματική, δημογραφική και ψηφιακή πρόκληση. Αν πραγματικά θέλουμε να μετασχηματίσουμε την Ευρώπη μα στην πρώτη ουδέτερη ήπειρο όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα πυλώνα και πόλο κόμβο καινοτομία και έρευνα και επιχειρηματικότητα, θα πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τι καλύτερε δυνατέ ε, δυνατότητε για τι επιχειρήσει μα και του οικονομικού μα παράγοντε. Και αυτό ακριβώ τονίζει άλλωστε και η συντάκτρια τη στο κείμενο τη αυτό. Καταθέτω μια σειρά από τροπολογίες κάπως τεχνικής φύσης και αναφέρομαι καταρχάς στο επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει και να πλαισιώσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Λέω ότι θα πρέπει μέσω της, ε, του πρασινίσματος οικονομίας να δημιουργηθούν νέες θέσεις, οικολογικές θέσεις απασχόλησης Λέμε επίση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισότητα στις ευκαιρίες απασχόλησης, να μειώσουμε τη φτώχεια και να αυξήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των διαφορετικών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αναλόμαστε σε περιττές συζητήσει για τους καθαρούς συνεισφέροντες και τους καθαρούς αποδέκτες. Νομίζω ότι Μόνο αν καταφέρουμε να έχουμε μία συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα καταφέρουμε να έχουμε μία πιο ενισχυμένη κοινωνική πτυχή στον προπολογισμό μα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε επίση να προωθήσουμε περισσότερο του κλιματικού μα στόχου. Θα πρέπει το νέο πολιτεύσιο νομοσυνομικό πλαίσιο να καλύπτει χρηματοδοτικά και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά και το μηχανισμό και το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση, κάτι το οποίο δεν το ανέφερε ρητά η προηγούμενη Φιλανδική Προεδρία και νομίζω ότι θα πρέπει ο νέος αυτός προπολογισμός και το ευρωπαϊκό εξάμεινο να μπορούν να καλύπτουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την οικολογική ενεργειακή μετάβαση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρέισεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη συντάκτρια της γνωμοδότηση. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε και εμείς όπως η ομάδα Renew να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθηθεί, αλλά επίσης και τα όσα θα πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπα προλαλήσαντας, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εργαστούμε στα πλαίσια ενός νέου οικονομικού μοντέλου και να τονίσουμε πραγματικά ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικέ αλλαγέ. Θα πρέπει δηλαδή να προσεγγίζουμε πλέον την οικονομία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε όλες τις πτυχές της, δηλαδή και την κοινωνική και την περιβαλλοντική πτυχή. Και αυτό συνδέεται λίγο και με την όλη συζήτηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν σε σχέση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τι θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του δημοσιονομικού κανονισμού και τι όχι. Ξέρετε ότι ήδη στις αρχές της εβδομάδας έγινε και μια συζήτηση μέσω διαφόρων άρθρων που δημοσιεύθηκαν στον τύπο. Για μας είναι σαφές ότι θα πρέπει τα πράγματα να αποσαφινιστούν και θα μπορούσε και αυτό να συμπεριληφθεί κάπως στη γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και με το μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί και αυτός ο σύσταση αυτή τη γνωμοδότηση. Στόχος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να συντονίσουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές και να αποφύγουμε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κυρία Μαρκέ, σωστά αναφέρετε στην έκθεσή σα την πρόκληση τη δημογραφική στην Ευρώπη. Και θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό για λίγο. Η δημογραφία στην Νότια Ευρώπη έχει αποτελματωθεί, διότι κάνουν ένα παιδί κυρίω εκεί και καταρρεί ανατολικά λόγω τη μετανάστευση εντό τη Ευρώπη. Κάποια στοιχεία. Η Ρουμανία έχασε ένα πέμπτο του πληθυσμού τη. Η Κροατία, η Βουλγαρία 5 με 10% από όταν μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για του νέου. Υπάρχει ή τη χρηματοδότηση να συντάξει και όχι μόνο. για τη χρηματοδότηση των συντάξεων και όχι μόνο. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και στα κράτη τη Βαλτική. Αυτή η διαφορά δημογραφική αυξάνει τι οικονομικέ διαφορέ, Υπάρχει κίνδυνο ανισορροπιών. Θα ήθελα να προσέξω ότι αυτή η δημογραφική μεταφορά, οι μεταφορέ οι μετακινήσει είναι οικονομικέ. Επενδύει 20 χρόνια, 25 χρόνια στη Ρουμανία το κράτο για κάποιον και πτώ πάει μεταναστεύει στη Γαλλία για να καλύψει την έλλειψη γιατρών στη Γαλλία είναι μεταφορά οικονομική από την Ανατολή προς τη Δύση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το brain drain μέσω των Ταμείων των Ευρωπαϊκών για να διορθωθεί η ανισορροπία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί τη Επιτροπή Προπολογισμών. Μπορούμε να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή είναι ένα σύστημα αντιστάθμιση. Ευχαριστώ την κυρία Μάρκε που έβαλε την δημογραφική πρόκληση στην έκθεσή τη και θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό. Θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το ε, σημείο μέσω τροπολογιών. Άλλα σχόλια. Κυρία Παπαδημούλη. Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο Μαρκές. I would like to thank Κόρικ Μαρκές for it. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τη συνάδελφο Μαρκές για το σχέδιο γνωμοδότησης που μας έστειλε. Ήδη έχουμε μια αλλαγή στον τίτλο από ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί στο μεταξύ έχει μπει στην ατζέντα και το Green New Deal. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει εκτός από τον τίτλο να δούμε, καθώς το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει μπει στο δέκατο κύκλο εφαρμογής του, και την ανάγκη επανασχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χρειαζόμαστε ένα ολιστικό σχέδιο για δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και πρέπει εκτός από το Green New Deal να δούμε ότι η μονόπλευρη προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε αριθμούς και λογιστικά μεγέθη με απουσία της κοινωνικής διάστασης έχει οξύνει επικίνδυνα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός της Ευρωζώνης κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η προηγούμενη συνάδελφος μόλις αναφέρθηκε σε μερικές από αυτές που έχουν σχέση με τη συνοχή και το brain drain. Άρα έχουμε σημάδια που μας επιβάλλουν ένα επανασχεδιασμό και αλλαγές. Η ίδια η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εργασιακή φτώχεια και οι εντυνόμενες ανισότητες. Είναι θετικό ότι στην γνωμοδότηση που μας παρουσίασε η συνάδελφος Μαρκές αναφέρεται στην ανάγκη να ξαναεστιάσουμε τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να τους συνδέσουμε με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε και πράγματα και προτεραιότητες. Με αυτήν την διάθεση θα καταθέσουμε ε, εκ μέρους της ομάδας μας και τροπολογίες μέσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τζόντσα. Ευχαριστώ. Α, με επιτρέψετε να μίσω πολωνικά. Μιλάμε ταυτόχρονα για πολλά πράγματα. Χαιρετίζουμε το ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ένωση σε διάφορους τομείς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως, πρέπει να πω ακόμη πως αυτό περί διαφορετικών σημείων εκκίνησης είναι εξίσου σημαντικό. Για τις διάφορες δράσεις υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες. Ένα παράδειγμα είναι ο κατώτατος μισθός. Εμείς είμαστε κατά για διάφορους λόγους. ή για άλλες προτάσεις, ε, παραδείγματο χάρη για τη φορολογία. για μια αρμόδια αρχή και αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος, όμως η ανάπτυξη σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθηθεί. Υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία αλλαγής, μετασχηματισμού των κρατών μελών. Το βλέπουμε και σε επίπεδο περιφερειών, αλλά και γενικά στο επίπεδο των κρατών μελών. Είναι τελείως διαφορετικά τα σημεία εκκίνησης. Πρέπει να δώσουμε έμφαση ε, στην έλλειψη αποκλεισμών και στη δίκαιη μετάβαση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ε, ε, λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες και χώρες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Πού βρίσκονται αυτές οι χώρες, έχουν καταφέρει να ευθυγραμμιστούν με τις υπόλοιπες ή υπάρχει υποβάθμιση. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα επιτόπου. Η δίκαιη μετάβαση είναι σίγουρα μια προτεραιότητα. Αλλά για να κρίνουμε τη δίκαιη μετάβαση πρέπει να δούμε τι κατάσταση ισχύει σε κάθε χώρα. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παναλαμβάνω όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει πραγματικότητα. Για να μην κάνουμε τελικά βήματα προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Κυρία Μάρκες, για να ολοκληρώσετε την συντομία παρακαλώ, γιατί χτυπάει ήδη την πόρτα μας ο κύριος Μάριτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις συνεισφορές τους. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι πρόκειται περί γνωμοδοτήσεως. Η Επιτροπή Οίκων έχει τον ε, κύριο ε, εισηγητή. Όπως σας είπα, ήθελα να υποβάλω κάποιες συστάσεις. Ως ήθιστε σε μια γνωμοδότηση, ε, πρέπει να προτείνουμε στον αρμόδιο εισηγητή της οίκων κάποια πράγματα. Αλλά για να είμαι σύντομη θέλω να πω το εξή. Πράγματι, παρόλο που πρόκειται περί γνωμοδότησης, μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Μας ενδιαφέρουν όλα. Υπάρχει δημοσιονομικός αντίκτυπος από όλα αυτά που συζητούμε. Αντίκτυπο τη Πράσινη Συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και για το θέμα των ίδιων πόρων. Ευχαριστώ όλου για τα σχόλιά του. Ακούστηκαν κάποιες προτάσεις για αλλαγέ που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην έκθεση για τροπολογίε. Η προθεσμία για τις τροπολογίε είναι 28 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ όλους σας για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις και τις τροπολογίες που προτείνατε στη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σημεία 10 και 11 θα συζητηθούν το απόγευμα. Μετά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων, επίσης θα ψηφίσουμε για το Πεκίνο. Να ξεκαθαρίσω ότι χρειάζομαστε απαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε τον κύριο, θα καλωσορίσω τον κύριο Μάριτς και θα συνεχίσουμε. Uh, Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Καλωσορίζω θερμά τον κύριο Τζάφκο Μάριτς. Όχι μόνο τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ και ειλικρινά που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ο κύριος Μάριτς είναι υπουργό Οικονομικών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σαν υπουργό Οικονομικών είναι για έξι μήνες τώρα και πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Αυτή η επίσκεψη αναμφισβήτητα είναι ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά το πνεύμα συνεργασίας της Κροατικής Προεδρίας για συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων για όλα τα θέματα και βέβαια και για τα θέματα που αποτελούν άμεσο αντικείμενο της Επιτροπής μας. Αρκετά σημαντικά θέματα που εμπίπτουν στην Επιτροπή προϋπολογισμών εκκρεμούν ή είναι θέματα που ανοίγουν τώρα επικρατικής προεδρίας, όπως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ίδιοι πόροι και τα σχετικά μέσα στον τομέα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, κράτος δικαίου, το νέο το επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και διαδικασία προς έγκριση του προϋπολογισμού του 2021. Βέβαια, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν είναι τα πάντα στην εντολή και στην αρμοδιότητα ΕΚΟΦΗΝ και η Κροατική Προεδρία πρέπει να έρθει σε επαφή και με τη Γερμανική Προεδρία όσον αφορά τον προπολογισμό του 2021 και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Κύριε Μάλιτς, προσβλέπουμε στις προτεραιότητες που παρουσιάσατε και τον σχεδιασμό της Κροατικής ε, Προεδρίας στους προαναφερθέντες τομείς. Με τα χαράς να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και να είμαι σε θέση να σας μιλήσω και να προβώ σε κάποια σχόλια, να κάνω κάποιες εναρκτήριες δηλώσεις από την πλευρά μας που είμαστε το νεότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη φορά που έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Έχουμε θετικά συναισθήματα γι' αυτό. Όσον αφορά την Προεδρία όμως, γνωρίζω πολύ καλά και εγώ ότι έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας μπροστά μας που ανέλαβαν πολλοί και στο Ζάγκρεμπ και στις Βρυξέλλες. Προσβλέπουμε στην Προεδρία μας. Χτες είχαμε την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου που την ηγεσία Κροάτη Υπουργού και πήγε καλά νομίζω. Μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Αυτό θα έλεγα. Αυτή είναι η, πρώτη μου η δεύτερη εμφάνισή μου σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, μίλησε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ μόλις τώρα και ζητώ συγγνώμη που επαναλαμβάνω πράγματα για σας που ήσασταν και σε εκείνη τη συνεδρίαση και τα ακούσατε. Τελειώσαμε τη συνεδρίασή μας εκεί, ήταν ε, αρκετά καλή όσον αφορά τη συζήτηση και ο πρόεδρος είπε ότι η ιδέα ήταν να απαντηθούν οι περισσότερες δυνατές ερωτήσεις, δυνατόν ερωτήσεις όσον αφορά τα σημαντικά θέματα αλλά όταν μιλάμε ως Προεδρία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προπολογισμό για τον επόμενο χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι στην αρχή είμαστε κάπως περιορισμένοι στον τομέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιμένουμε πολιτικούς προσανατολισμούς για τα διάφορα θέματα. Χαίρομαι που θέσαμε κάποια ζητήματα και για μένα θα ήταν πολύτιμο να συλλέξουμε ερωτήσεις και σχόλια από σας, από την Επιτροπή σας. Να κάνω σύντομη παρουσίαση όσον αφορά τι δημοσιονομικέ προτεραιότητε και τον προπολογισμό από πλευρά κρατική προεδρία και μετά από αυτό μπορούμε να πάμε στι ερωτήσει και τι απαντήσει. Ζούμε σε ενδιαφέρουσα εποχή. Όταν λέω ενδιαφέρουσα, ε, είναι κάτι σχετικό ενδιαφέρουσα περίοδο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε ένα νέο θεσμικό κύκλο και θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Προεδρία μα, με τη βοήθεια των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έλεγα. Είναι σημαντικό εγχείρημα. Το σύνθημά μας είναι ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο με προκλήσεις. Αυτό μπορεί εύκολα να μεταφραστεί στις παρούσες περιστάσεις και ενελοποιηθεί. Ναι, οι ευρωπαϊκοί κύκλοι ξεκίνησαν και εμείς σαν Προεδρία θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι μόνο καλά, αλλά επικοδομητικά με σωστή προσέγγιση, θετικά αποτελέσματα, ελπίζουμε στο τέλος της Προεδρίας μας. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Τέσσερις βασικές προτεραιότητες έχουμε, όμως παράλληλα ή αλληλένδετες είναι και άλλες. Κάποια θέματα που θέλουμε να θέσουμε, που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Να ξεκινήσω από τις γενικές προτεραιότητες. Πρώτα, θέλουμε αναπτυσσόμενη Ευρώπη. Θέλουμε ισόρροπη, βιώσιμη, συμπεριληπτική ανάπτυξη στην Ευρώπη οικονομική και αντιμετωπίσουμε και τα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης. Θα ζητήσουμε μια ισχυρή ενιαία αγορά, αύξηση ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω συνοχής και σύγκλησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζοντας το πιεστικό πρόβλημα του κλίματο. Σχετικά με αυτό, θέμα θα ξεκινήσουμε οριζόντιε συζήτηση όσον αφορά τη νέα πράσινη συμφωνία για την Ευρώπη. Δεύτερη προτεραιότητα, η Ευρώπη που συνδέει. Να προωθήσουμε πρωτοβουλίε που συμβάλλουν στι μεταφορέ, την ενέργεια και ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, αντιμετωπίζοντα και τα προβλήματα που δημιουργεί η ψηφιοποίηση και η νέα τεχνολογία. Επίσης θα θέλουμε να προωθήσουμε και άλλες πρωτοβουλίες για ισχυρότερε διασυνδέσει μεταξύ των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μέσω αθλητισμού, πολιτισμού, παιδεία κλπ. Τρίτη προτεραιότητα είναι η Ευρώπη που προστατεύει ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών εσωτερικά και εξωτερικά. Θα επεξεργαστούμε ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση. Νέα στρατηγική κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον χώρο ελευθερίας ε, δικαιοσύνης και δικαιοσύνης. Μετά θέλουμε μια Ευρώπη που έχει επιρροή, που ηγείται και στον κόσμο και στη γειτονιά. Οπότε θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ Δυτικά Βαλκάνια το Μάιο του 2020 και τη Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική Γειτονιά επίσης. Θέλουμε, ξέρουμε ότι η προσχώρηση και ένταξη μεταλλάσσει καταστάσεις και θέλουμε να παρόλα αυτά να πληρών, όταν πληρούνται τα κριτήρια για ένταξη να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Χρειαζόμαστε και οικονομική υποστήριξη για όλα αυτά στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ή εντό του προπολογισμού θέλουμε να κινηθούμε το ετησίου. Το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, το πακέτο με όλε σχετικέ προτάσει είναι προτεραιότητα για μα, ύψιστη προτεραιότητα τη Προεδρία. Όπω ξέρετε, η διαδικασία όμω είναι στα χέρια του Προέδρου του Συμβουλίου, του κ. Σαλ και ο ρόλος της κρατικής προεδρίας σε αυτό το τομέα είναι περιορισμένος. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο σε τομεακέ νομοθετικέ προτάσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να επιτρέψουμε ομαλή μετάβαση μεταξύ τη παρούσα γενιά των προγραμμάτων και των μελλοντικών. Σχετικά με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, εμεί, σαν Προεδρία, ε, θέλουμε να οικοδομήσουμε ισχυρέ σχέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε τι καθιερωθήσει πρακτικέ ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο πριν και μετά το συμβούλιο, τα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων όταν θα είναι στο, στο πρόγραμμα η συζήτηση το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πολύ σημαντική τη συνεργασία μας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Από τη στιγμή που θα έχουμε λάβει προσανατολισμού από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κροατική Προεδρία επίση θα ξεκινήσει τη τελική φάση της κατάρθρων εξετάσεως των νομοθετικών προτάσεων που θα αποτελέσουν το πακέτο για τους ίδιου ε, πόρους. Όσον αφορά τη διαδικασία του ετησίου προπολογισμού, ο προπολογισμό για το 2021 θα είναι ε, το πρώτο σημείο στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο προετοιμάζει τώρα κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2021 και θα παρουσιαστούν στου εκπροσώπου αυτή τη Επιτροπή ε, στον τριμερή διάλογο τη Άνοιξη. Η ετήσια διαδικασία μετά θα ξεκινήσει κανονικά από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσει για το σχέδιο προπολογισμού. Οι εργασίε από πλευρά Συμβουλίου θα ακολουθήσουν την ηγεσία της μελλοντική γερμανικής προεδρίας. Επίσης θα ήθελα ακροθυγουχώς να αναφερθώ στον τομέα των νομοθετικών φακέλων που θα σας ενδιαφέρουν. Έχοντας προσανατολισμούς από το Eurogroup, στις 9 Οκτωβρίου το Συμβούλιο επεξεργάστηκε τη μεταρρύθμιση, τα προγράμματα μεταρρύθμισης και υποστήριξης. Η προηγούμενη Προεδρία μοιράστηκε το κείμενο με σας Παρόλο που σε αυτή τη φάση δεν είναι επίσημη θέση του Συμβουλίου, τα βασικά οικοδομικά στοιχεία υπάρχουν. Σαν Προεδρία πιστεύουμε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να βασιστεί στα οικοδομικά, τα δομικά αυτά υλικά. Σημαντικά θα προωθήσουν αυτά τις εργασίες των συνομοθετών, αλλά και θα εξοπλίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα σωστά εργαλεία που θα υποστηρίζουν τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις Είχαμε διεξοδικότατη συζήτηση στην προηγούμενη Επιτροπή περί της κατεπίγουσας ανάγκης για ευαισθητοποίηση σχετικά με την τόνωση και βελτίωση και αύξηση της ε, ε ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Και συμπεράσματα πλευράς Ευρωβουλευτών και από Προεδρίας ε, ήταν σαφέστατα, θα έλεγα, ότι η υποστήριξη και οποιοδήποτε στοιχείο τόνωσης διαθωτικών μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτά που απαιτούνται και με το παραπάνω. Όσον αφορά την το πρόγραμμα για υποστήριξη για μεταρρυθμίσει, να υποστηρίξω τις σημαντικότερες, να αναφέρω τις σημαντικότερες αλλαγές όμω που γίνονται εν συγκρίση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έχουμε από τη μια πλευρά εργαλεία για τις μεταρρυθμίσεις αντικαθίσταται με ένα κεφάλαιο που καθορίζει το δημοσιονομικό μέσο για ανταγωνιστικότητα και σύγκληση για την Ευρωζώνη. Δεύτερο, εργαλείο μεταρρύθμιση σύγκληση για τι χώρε εκτό ευρωζώνη δημιουργήθηκε και καθιστά το μέσο σύγκληση και τέλο, μικροαλλαγέ έχουν γίνει όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη και το σχετικό εργαλείο. Καλωσορίζουμε το μνημόνιο συνεννόηση που επετεύθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα οικονομικά μέσα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα Invest EU και θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο επ' αυτού εάν τελικά επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτές είναι πρώιμες ημέρες της ε, Προεδρίας μας, πρώτες ημέρες. Φιλοδοξία μας είναι να επιτευχθεί οικονομική πρόοδος όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα το επόμενο εξάμεινο και ελπίζουμε αυτό να το πετύχουμε σε επικοδομητικό πνεύμα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ ολοκληρώνω την περιγραφή μου και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάριτς για τα εισαγωγικά σας αυτά λόγια. Λοιπόν, πώς θα κινηθούμε τώρα από εδώ και πέρα. Εγώ σας προτείνω καταρχάς να πάρουν το λόγο οι συντονιστές της Επιτροπής μας και αν το επιτρέψει ο χρόνος, γιατί μπορούμε να πάμε μόνο μέχρι τη μία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye για τους υπόλοιπους ομιλητές στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο συντονιστή, τον κύριο Φερνάντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Δημοκρατίας της Κροατίας και Υπουργό Οικονομικών, είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε στα πλαίσια μιας αγαστής εταιρική σχέσης. Η συνοχή αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο, η σύγκληση επίσης, το πολιτές νομικό πλαίσιο επίσης. Θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι όντως θα έχουμε την κατάλληλη βέλτιστη συμφωνία όσον αφορά το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα καταφέρουμε όμω να πετύχουμε μια συμφωνία αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και νέου ιδίου πόρου. Εμένουμε στο στοιχείο αυτό και θα χρειαστούμε βέβαια και μια μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Εσείς τι ρόλο θα διδραματίσετε στην όλη αυτή διαδικασία προκειμένου δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατό. Και ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρείτε ότι ακολουθήσαμε τη σωστή μεθοδολογία. Εμείς μιλάμε για 1,3% όσον αφορά το καθάριστο εθνικό εισόδημα. Αυτό το 1,3% δεν είναι βέβαια ένα τυχαίο ποσοστό. Το ποσοστό αυτό διέκοψε το μικρόφωνο το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στα κονδύλια τα οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα προγράμματα αυτά χρειαζόμαστε ένα καλό περιεχόμενο και θα πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να έχουμε περικοπές στην έρευνα, τη συνοχή, τη σύγκληση. Και έχουμε και μία άλλη βασική αρχή την οποία ακολουθούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επί τη οποία θα ήθελα και τη δική σα την άποψη. Οι νέε πολιτικέ χρειάζονται φρέσκο χρήμα, φρέσκια χρηματοδότηση. Νέα προγράμματα και νέε προτεραιότητε θα πρέπει να έχουν επιπρόσθετα κονδύλια, επιπρόσθετη νέα χρηματοδότηση. και ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά το δημοσιονομικό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση. Με τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή το εργαλείο αυτό φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τις πλούσιες χώρες και όχι τις πιο ευάλωτε αυτέ οι οποίε θα πρέπει να συγκλίνουν προ τι υπόλοιπε. Σε κάθε περίπτωση πάντως κύριε Υπουργέ μπορείτε να βασίζεστε στη δική μα υποστήριξη και να καταλήξουμε σε μια γρήγορη συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και θέλω να ελπίζω ότι θα υποστηρίξετε και την πρόταση αλλά και τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα το ποσοστό το οποίο εμεί προτείνουμε για τη χρηματοδότηση 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματο. Αυτό δεν αποτελεί απλώ ευσεβή πόθο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά μια πραγματικότητα και να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω την Κροατική Προεδρία. Δεν παρακολούθησα τη συζήτηση που έγινε στην ΕΚΟΝ, αλλά ο συνεισηγητής για το πρόγραμμα που των επενδύσεων η εισηγητρία έκανε κάποιες ερωτήσεις και εγώ θα πω αντίστοιχα πράγματα διότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και με αυτό και με άλλους μηχανισμούς. Πρώτον, διότι Υπήρξε παράλυση στο Κοινοβούλιο γιατί περιμέναμε να δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις ε, στο Eurogroup δεν θεωρήσαμε ότι είχε νόημα εμείς να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε την ε, πρόταση της Κομισιόν όταν ε, θα περιμέναμε διαφορετικά πράγματα σχετικά τουλάχιστον από το Συμβούλιο και το Eurogroup. Άρα είχαμε κάπως παραλύσει. Επίσης το πρόγραμμα αυτό εξαρτάται απόλυτα από τις διαπραγματεύσεις πάνω στο πει και σε ό,τι αφορά τα ποσά που δεν θα είναι τα ίδια το να έχουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων στήριξη των μεταρρυθμίσεων 10-15-25 ε, ε, και τα ποσά, τα κριτήρια, οι προτεραιότητες ανάλογα με το ποσό θα διαφέρουν. Και επίσης Όταν γίνεται ε, σε αυτό το πρόγραμμα αναφορά, ε, στο διαπραγματευτικό κουτί, ουσιαστικά περιλαμβάνονται κάποια βασικά σημεία, τα οποία θα είναι αντικείμενα διαπραγμάτευση μεταξύ Συμφωλίου και Κοινοβουλίου. Άρα, το Κοινοβούλιο ε, τι διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει. Δεν ξέρουμε τα ποσά δεν ξέρουμε ποια είναι τα βασικά σημεία για την κατανομή, για τη χρήση, για τα κριτήρια που είναι σε αυτό το nego box, στο διαπραγματευτικό κουτί και πρέπει να αποφασίσει με ομοφωνία το Συμβούλιο. Πώ θα τα αντιμετωπίσει, πώ θα αντιμετωπίσετε αυτέ τι διαπραγματεύσει στο Κοινοβούλιο. Και έχουμε και μια ακόμη ε, συνιστόσα που, περιπλέκει τα πράγματα. Ε, τομεακές εκθέσεις ε, θα είναι από την Προεδρία ε, και άλλα θέματα από τον κύριο Μισελ. Άρα πώς εμείς μπορούμε να ε, προσεγγίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσει ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Αγιέ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψε. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσει, για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, τα τελευταία νέα είναι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για πάγωμα των διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο. Και θα ήθελα να μου πείτε η Κροατική Προεδρία πώς θα αντιδράσει σε αυτή την ισχυρή απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Θα επιταχύνετε εσείς τις συζητήσεις σε τομεακό επίπεδο μια από τι τελευταίε πιο πρόσφατε εξελίξει μετά από αυτή την απόφαση ήταν η απόφαση τη Επιτροπή Ρέγγι από χθε να παγώσει τι συζητήσει για την πολιτική συνοχή. Και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα. πολιτική συνοχή ε, είναι προσφυλής ιδιαίτερα στην Κροατία και γι' αυτό η θέση της Κροατίας ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό και με τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Και γι' αυτό το θέμα, όσο και για άλλες, όσο έχετε ένα σύμμαχο στο πλευρό του Κοινοβουλίου. Πώς λοιπόν θα μας αξιοποιήσετε, πώς θα μας χρησιμοποιήσετε εσείς, εμάς, το Κοινοβούλιο, του Ευρωβουλευτές, για τις θέσεις που θέλετε να παρασπιστείτε πιο έτσι προσωπικά ως κρατός μέλος. Τρίτο ερώτημα, ήδη οι πόροι. Στο πρόγραμμα εργασίας σας λέτε πως ε, θα εστιάσετε στην ε, λήξη των ε, συζητήσεων και των για τους ίδιους πόρους, στην οριστικοποίηση. Δηλαδή αυτό τι θα πει. Θα το δείτε στο ίδιο επίπεδο με τις δαπάνες, το θέμα αυτό. Και πότε θα λήξουν αυτές τις πραγματεύσεις. Κάτι άλλο. Η μεταρρύθμιση των ιδιών πόρων. Ξέρετε και το είπαμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Ποια είναι απόψεις σας από αυτού. Και για την κρατική προεδρία και το πρόγραμμα της κάτι τελευταίο λέτε ότι θέλετε δίκαιη φορολογία με προσαρμογή των φορολογικών κανόνων στην ψηφιοποίηση οικονομίας και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο ρόλος του ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού ε, σε έσοδα και δαπάνες ποιος είναι κατά την άποψή σας Πιστεύω θα μπορέσετε να πείσετε τους πλέον απρόθυμους ε, συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σάντρισεν. Σας ευχαριστώ κύριε Μάριτς. Εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως ότι είστε εδώ παρόν σήμερα στην Επιτροπή μας και θεωρούμε ότι μπορείτε πραγματικά να δραματίσετε ένα σημαντικότατο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα και ιδίω για τα τομεακά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ο ρόλος σας θα είναι πολύ σημαντικός και χρειάστηκε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε και με άλλες χώρες στο παρελθόν. Η δική σας η χώρα πάντως είναι πολύ σημαντική, διότι ε, Ξέρω ότι ε, είχατε υιοθετήσει ε, διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν σε σχέση δηλαδή με τις χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς και παλαιότερα είχαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εσείς μπορείτε να φωτίσετε μια διαφορετική πλευρά των πραγμάτων. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που κάνουμε την όλη αυτή συζήτηση, η οποία δεν θα πρέπει να έχει να κάνει μόνο με αριθμητικά δεδομένα, αλλά και με ουσιαστικέ αξίε. Θα ήθελα να θέσω ένα διαφορετικό λοιπόν ζήτημα να αναφερθώ σε μία από τι προτεραιότητές σας. Πριν από λίγο είπατε ότι θέλετε να προστατεύσετε την Ευρώπη, ότι αυτό αποτελεί μία μια προτεραιοτητα σας. Και είπατε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί και με το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών. Ακούσαμε ότι στα εξωτερικά σύνορα της Κροατίας υπήρξαν αναγκαστικές επαναπροωθήσεις, επιστροφές μεταναστών. Ξέρουμε ότι ε, πολλά κοινοτικά κονδύλια δαπανώνται για την προστασία των εξωτερικών αυτών συνόρων και της δικής σας της χώρας λοιπόν. Συμφωνείτε λοιπόν ότι ο προπολογισμό μα θα πρέπει να, να κάνει και με σημαντικέ αξίε και ότι θα πρέπει να προασπιστούμε και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όταν δαπανούμε κοινοτικά κονδύλια. Και τι έχετε να πείτε για τι διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε αναφέρονται σε μια πολύ δεινή κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τη Κροατία. Ξέρετε ότι ε, τα όσα θα μας πείτε θα επηρεάσουν ε, και τις διαπραγματεύσει που θα κάνουμε για την μεταναστευτική πτυχή του κοινωνικού προπολογισμού. Σας ευχαριστούμε κυρία Λαπόρτ, έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην Επιτροπή μα και μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου παρουσιάσετε το πρόγραμμά σα. Δύο ερωτήσει λοιπόν. Η πρώτη έχει να κάνει με του ιδίου πόρου. Αποτελούν από ό,τι φαίνεται προτεραιότητε κρατική προεδρία. Η πολιτική μου ομάδα, η ID, είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστική σε σχέση με τους ιδίους αυτούς πόρους και τη σχετική τους μεταρρύθμιση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, οι ίδιοι αυτοί οι πόροι φαίνεται ότι θα λειτουργήσουν εις βάρος των καθαρών συνεισφορών που γίνονται από τα κράτη-μέλη. Ενδεχομένως λοιπόν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από τα κράτη-μέλη κατά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτο ερώτημα αυτό. Δεύτερον, η διαπραγμάτευση του μελλοντικού πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2027. Μεγάλες οι αποκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλουν να έχουν ένα πιο ουσιαστικό προπολογισμό, ενώ το Συμβούλιο θέλει να κάνει συνεχείς περικοπές και από ό,τι φαίνεται δεν προωθεί έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό προπολογισμό. Ποια θα είναι η δική σας συστάση και πώ προβλέπετε τη μελλοντική εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζόντσα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Είστε όντω από τι πιο νέε, η πιο νέα μάλλον χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι θετικό γιατί θα καταφέρετε όντω να έχετε μια φρέσκια ματιά, φαντάζομαι, σε σχέση με διάφορε πολιτικέ. Θεωρώ λοιπόν ή θέλω να ελπίζω ότι η συμβολή της Κροατίας θα είναι αποτελεσματική και ουσιαστική. Μας παρουσιάσατε τέσσερις τομείς ως βασικές σας προτεραιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το ακόλουθο. Στα πλαίσια των προγραμμάτων που μας παρουσιάσατε, προβλέψατε να ασχοληθείτε με το βασικό αυτό σχέδιο που είχε να κάνει με τις τρεις θάλασσες κατά τη διάρκεια της κρατικής προεδρίας. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τις σχετικές αυτές πρωτοβουλίες και να έχετε μια χρηματοδότηση βασικά ουσιαστική για την πολιτική αυτή. Έπειτα, όσον αφορά τα Καρπάθια, η Κροατία εν μέρη καλύπτει και την περιοχή αυτή. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι η χρηματοδότηση που προβλέπεται όσον αφορά τι διασυνοριακέ ζώνε και τα σχετικά διασυνοριακά προγράμματα για την περιοχή των Καρπαθίων. Οι πολιτικέ αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ξέρετε, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε πραγματικά μια ισχυρή ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε λοιπόν τα διασυνοριακά αυτά προγράμματα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, ο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Μάριτς, ε, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Κροατική Προεδρία, αλλά θέλω να προσθέσω και το αυτονόητο ότι το πόσο πετυχημένη θα είναι η Προεδρία σας θα εξαρτηθεί πρώτον από το αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου και από το πόσο εσείς θα διεκδικήσετε φιλόδοξους στόχους που να τους πετύχετε ξεκινώ από το θέμα της συνοχής. Ο κύριος Πλένκοβιτς πριν λίγες ημέρες παρουσιάζοντας τους στόχους της Κροατικής Προεδρίας έβαλε πολύ ψηλά το θέμα της συνοχής. Και σωστά. Η προτεραιότητα όμως που θέτει η Κροατική Προεδρία ακυρώνεται από τις προτάσεις που έχει καταθέσει μέχρι τώρα το Συμβούλιο όπως μας τις παρουσίασε η προηγούμενη Προεδρία, η Φιλανδική. Και επειδή είστε και υπουργό Οικονομικών εκτός από αναπληρωτής Πρωθυπουργό, σας μιλώ με αριθμούς. Η πρόταση που υπάρχει σήμερα στο τραπέζι από το Συμβούλιο προβλέπει μείωση των κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή 13%. Ειδικά για το Ταμείο της Συνοχής προβλέπει μείωση 47% και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο περίπου μείωση 10%. Είναι αδύνατον πιστεύω να κάνει κανείς περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύεται αυτή την αντίφαση ανάμεσα στους στόχους της Κροατικής Προεδρίας και στις μέχρι τώρα προτάσεις του Συμβουλίου να τη γεφυρώσετε. Το δεύτερο αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που κομμάτι του είναι και ο προϋπολογισμός του 2021. Εδώ η κατάσταση βρίσκεται σε τέλμα διότι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου όπως παρουσιάστηκαν από τους συντονιστές και των άλλων πολιτικών ομάδων για 1,3% του ΑΕΠ προκύπτουν από τους στόχους που έχει θέσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτά τα χρήματα χρειάζονται για να πετύχουμε τους στόχους. Δεν είναι μια αυθαίρετη κατασκευή. Και η, απόσταση ανάμεσα στην πρόταση του Συμβουλίου και στην πρόταση του Κοινοβουλίου είναι πολύ μεγάλη. Ήταν απογοητευτική η πρόταση Φιλανδικής Προεδρίας. Πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που είχε το, το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σε αριθμούς απέχει η πρόταση του Συμβουλίου η ισχύουσα 236 ευρώ από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι και μειωμένη κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την ισχνή κατά τη γνώμη μας πρόταση της Κομισιόν. Η ερώτησή μου σε αυτό το θέμα είναι ποιον ακριβώς ρόλο θα παίξει η Κροατική Προεδρία. Γιατί στο θέμα αυτό έχει μια εντολή και ο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, θα ασχοληθείτε ενεργά με αυτό το θέμα. Και επίσης ή θα το αφήσετε στον κύριο Μισελ. Και το δεύτερο, σκοπεύετε να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος στη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας ή θα είναι η Προεδρία σας μια Προεδρία Transit για να πάει το θέμα στην Γερμανική Προεδρία. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε και τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch για να μπορέσει μετά ο κύριος Μάριτς να απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις που το ετέθησαν. Ο κύριος Ρέσλερ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω κροατικά αυτή τη φορά. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Μάριτς. Καταρχάς ε, θέλω να σας ε, συγχαρώ που αναλάβατε την Προεδρία και για το καλό ξεκίνημα. Σίγουρα υπάρχουν πολλέ άλλες προτεραιότητε, αλλά οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ θα είναι ένα ζήτημα κλειδί για τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως η Κροατία θα έχει να παίξει σίγουρα κάποιο ρόλο ε, στη διάρκεια αυτή της Προεδρίας. Και αυτό κυρίως γιατί ο στόχος της συνοχής και των σχετικών κονδυλίων είναι να υπάρχουν επαρκείς ε, πρόδια ε, πόροι για τον παραδοσιακό πυλώνα της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της σημερινής εποχής. Τα ποσά που θα ενταχθούν στο ΠΔΠ ναι θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ξέρουμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα όλα μεταξύ τους, ο ένας τομέας με τον άλλον. Ακούσαμε πολλούς να μιλούν για το 1,3% του ΑΕΠ. Δεν το βγάλαμε από το μυαλό μας, ούτε έπεσε από τον ουρανό αυτό το νούμερο. Αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Έτσι μεταφράζονται σε αυτό το ποσό αν θέλουμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Δεν βλέπω λόγο να μην έχουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους στόχους, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τους πετύχουμε αν δεν υπάρξει και μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδιών πόρων. Προσωπικά λοιπόν θα με ενδιέφερε να μου πείτε ποια είναι η πρόοδος της μεταρρύθμισης. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το εξάμεινο αυτό, παράλληλα και με τις επραγματεύσεις για το ΠΔΠ και τα άλλα θέματα που θα σας απασχολήσουν. Σας εύχομαι να έχετε ένα επιτυχημένο εξάμεινο και ελπίζω να συνεργαστείτε στενά με το Ευρωκοινοβούλιο για να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν και το ΠΔΠ. Ευχαριστώ κύριο Λεβαντόφσκι. Συγχαρητήρια για την Προεδρία που αναλαμβάνετε κύριε Υπουργέ. Σίγουρο ο πραγματικός πανοκέφαλος είναι η Συμφωνία για το ΠΔΛΤΑΠΗ. Αλλά ευτυχώς δεν θα είναι πονοκέφαλο για την εκπεριτροπή στη Κροατική Προεδρία. Αλλά μάλλον θα είναι πλήρης ευθύνη του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Θυμάμαι την τελευταία φορά τον πρόεδρο Χέρμαν Φονορομπάι, ο οποίος ήταν ε, ε, αυτός που αναλάβει την πλήρη ευθύνη και κρατούσε στα χέρια του το πιδάλιο και δοκίμαζε και τις ε, αντοχές των πρωτευουσών, κατέβαζε νούμερα για να πάρει στο πλευρό του τον κύριο Κάμερον και τελικά ε, έκανε δώρα ε, στις κυβερνήσεις που δεν ήταν ε, ικανοποιημένε. Ελπίζω να έχει επίγνωση των ευθυνών το κύριο Μισελ, αλλιώς δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε συμφωνία διακυβερνητική. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση για το Κοινοβούλιο σε μια τέτοια περίπτωση. Σίγουρα η δική σας συμβολή γιατί είστε μια χώρα συνοχής θα είναι μεγάλη αλλά κατάρτιση ετήσιου προπολισμού χωρίς το πιδελταπή και αυτό θα είναι ένα άκρος ενδιαφέρον εγχείρημα. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς και εγώ τον Υπουργό για την διαθεσιμότητά του, για το ότι ήρθε να μας μιλήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Ξέρω ότι πήγατε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, όπως μας είπατε. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά ήρθατε εδώ στη δική μας Επιτροπή τώρα και ελπίζω ότι η παρουσία σας εδώ σήμερα θα αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον, για το πώς δηλαδή προτίθεται να συνεργαστεί στο μέλλον η Κροατική Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αναφέρομαι όλος ιδιαίτερο σε ένα ζήτημα το οποίο μας προκαλεί ανησυχία εδώ στην Επιτροπή Προεπολογισμών. και αναφέρομαι βέβαια στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, για το οποίο είμαι εισηγήτρια. Ελπίζω ότι η Κροατική Προεδρία θα συνομιλήσει με την ομάδα των φίλων της Συνοχής στη Λισαβόνα το Φεβρουάριο όταν θα γίνει εκεί μια συνάντηση προκειμένου πραγματικά να καταλάβει να συνειδητοποιήσετε τη σημασία της πολιτικής συνοχής και τη σημασία που θα έχει η πολιτική συνοχής για το επερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι στην συνάντηση αυτή του Φεβρουαρίου θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια πιο ευρή αντίληψη και εικόνα των πραγμάτων και θα καταφέρετε κατά αυτόν τον τρόπο να προσδώσετε ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας στι επερχόμενε διαπραγματεύσει. Κάποιες ερωτήσεις τώρα. Το λεγόμενο Nego το πλαίσιο διαπραγματεύση. Η Φιλανδική Προεδρία είναι αυτή η οποία δημιούργησε το πλαίσιο αυτό διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε τι δικέ του προτάσει και συστάσει, προσπαθώντα να διασφαλίσει ότι θα συμπεριληφθούν οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και όσον αφορά τι επιμέρου τομεακέ πολιτικέ και προτεραιότητε κάθε επιτροπή μα. Θέλουμε κατά αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι οι προτεραιότητε αυτέ θα συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά που τον Nego αναφέρεται σε διαδικασία συναπόφαση. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε, θεωρώ πολύ καλά την όλη αυτή η κατάσταση, γιατί προετοιμαζόμενους για τη σημερινή, σας, τη σημερινή μας συνάντηση, φαντάζομαι ότι θα μελετήσατε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω λοιπόν να σας κάνω την ακόλουθη ερώτηση. Η Κροατική Προεδρία προτίθεται να διατηρήσει το εφιστάμενο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, το εφιστάμενο Negobox, ή θα το μεταρρυθμίσετε. Δεύτερον, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο προλαλής σας ήδη σα έθεσε το ερώτημα αυτό. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργό σα στην Ολομέλεια μα είπε ότι θέλει να εγκρίνει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια τη κρατική προεδρία. Δεν θα μπορούσε να πει βέβαια και τίποτα άλλο ο Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να γνωρίσουμε και τη δική σα αξιολόγηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Τι πιστεύετε ότι μπορεί όντω να γίνει κατά τη διάρκεια τη κρατική προεδρία. Εν κατακλείδη, εύχομαι καλή επιτυχία στην προεδρία σα. Προφανώ επηρεάσει και το δικό μα το έργο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Όλμπρεχτ, έχει το λόγο. Και εγώ όπως οι συνάδελφοί μου θα μιλήσω σαν συνεισηγητής για το ποτέ δημοσιονομικό πλαίσιο όσα συσχετίζονται για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύσκολα θέματα. Ελπίζω η Προεδρία να πάει πολύ καλά, να υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με την Προεδρία. Κάτι που δεν ίσχυε στην προηγούμενη Προεδρία. Συμβολικά μας αντιμετώπισε η προηγούμενη Προεδρία με διπλωματικό τρόπο και μόνο. Και μας αγνόησαν τελείως θα μπορούσαμε να πούμε. Ελπίζω η Κροατική Προεδρία να παρουσιάσει διαφορετική προσέγγιση εναντί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει ότι έχετε κάπως διαφορετική προσέγγιση. Καλό σημάδι. Αυτό είναι το ένα. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι πιστεύουμε ότι πριν τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ομόφωνη απόφαση είναι αναγκαίο να γίνει δουλειά με το Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να περιμένουμε απλώς για ομόφωνη απόφαση. Μέχρι τότε θα είναι αργά. Θέλουμε να έχουμε πληροφορίες εκ των προτέρων είναι σαφές μήνυμα αυτό. Δεν θέλουμε να, να παρακολουθούμε από το περιθώριο τη διαδικασία. Θέλουμε να συμμετάσχουμε από την αρχή. Αυτό που είπαν συνάδελφοι πριν. Αναφερθήκατε, είπατε ότι η αρμοδιότητά μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι περιορισμένη. Ε, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Αν ο κύριος Μισελ λάβει απόφαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αν είναι υπεύθυνο για, τον... για τον Ego Box, για τι διαπραγματεύσει. Εσεί, σαν Προεδρία, είσαστε υπεύθυνοι για τομεακά ζητήματα. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν οι Ευρωβουλευτέ για τομεακά ζητήματα, σε εσά ή στον κύριο Μισελ. Διότι θα γίνονται παράλληλε εργασίε. Με τον κύριο Βαν Ρόμπο είχαμε κάποια εμπειρία, ήταν εντελώ διαφορετική κατάσταση και η πραγματικότητα. Ήταν πολύ παλιά, διαφορετικό κοινοβούλιο. Αυτό το κοινοβούλιο μαθαίνει. Και θέλει αυτό το κοινοβούλιο να γνωρίζει σε ποιον πρέπει να απευθύνεται. Ποιος είναι ο συνομιλητής μας. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη. Να γίνει επιμερισμός εργασιών. Ποιο είναι ποιο, ποιο κάνει τι. Αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μορεσάν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο στην Επιτροπή Προπολογισμών. Καταρχά να σα συγχαρώ επί της διαχειρίσεως της κρατικής οικονομίας, σταθεροποίησατε την ανάπτυξη, μειώσατε την ανεργία και μειώσατε και το δημόσιο χρέος. Στόχος σας να μπείτε στο μηχανισμό ισοτιμιών μέχρι το τέλος του έτους, καθοδόν προς την Ευρωζώνη. Είσαστε υπόδειγμα για πολλές οικονομίες που δεν είναι ακόμα στην Ευρωζώνη, συγχαρητήρια. Το θέμα μου τώρα, κύριε Υπουργέ. Ο ετήσιος προπολογισμός. Εσείς σαν Προεδρία το πρώτο εξάμεινο, του πρώτου εξαμήνου έχετε σημαντικότατο ρόλο. Μπορείτε να επηρεάσετε θετικά τον προπολογισμό. Γιατί το λέω αυτό. Κατά τη διάρκεια σα, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει του πολιτικού προσανατολισμού για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου. Έχετε δυνατότητα να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού τι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ω προτεραιότητε. Σε προηγούμενα χρόνια, πολύ συχνά, οι γραμματείε αντέγραφαν έγγραφα από χρόνο σε χρόνο. Οι Προτεραιότητε ήταν ε, ασφάλεια, ανάπτυξη κλπ. Καλά ακουγόταν οι προτεραιότητε. Το πρόβλημα ποιο ήταν. Τα λόγια των πολιτικών καθευτήριων γραμμών έδειχναν ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερο για την ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά όταν φτάναμε στα αριθμητικά στοιχεία, οι προεδρίες περιέκοπταν τα ποσά κυρίω τα κονδύλια που θα είχαν αντίκτυπο για την ανάπτυξη. Λέτε θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, αυτό λέγαμε, και μετά το Συμβούλιο πρότεινε περικοπε των ποσών, κυρίω για τον ορίζοντα 2020, για τα προγράμματα υποδομών και Λέγαμε θέλουμε να υποστηρίξουμε την ασφάλεια, στα λόγια, στην πράξη όμω είχαμε περικοπές στον αφορά το Ταμείο για τη Μετανάστευση. Και βλέπω μια ευκαιρία τώρα για πολιτική παρουσία τη προεδρία. Πώ θα την αντιμετωπίσετε, πώ προτίθεστε να κάνετε ευέλτιστη χρήση του σημαντικού αυτού βήματο που έχετε στη διαδικασία του προπολογισμού, να καθορίσετε πολιτικού προσανατολισμούς και να εξασφαλίσετε ότι δεν θα παραμείνουν κενά λόγια οι προτεραιότητες, αλλά έχουν πραγματικό αντίκτυπο όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό. Και μπορείτε να επηρεάσετε ε, και τι προτεραιότητε μέσω των προτεραιοτήτων σα και το υπόλοιπο τέτου. Όπω ρώτησε ο κ. Λεβαντόφσκι και εγώ θέλω να ρωτήσω πώ θα προχωρήσετε για τον ετήσιο προπολογισμό στο βαθμό που δεν έχουμε ακόμα συμφωνία όσον αφορά ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπονφρίσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, και εγώ σας επιθυμώ τις καλύτερες μου ευχές και ελπίζω να ξεκινήσετε σύντομα τη δουλειά σας και να μην σας κάνετε να χάνετε πολύτιμο χρόνο οι ερωτήσεις μας, αλλά να μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Εν ονόματι της φιλίας Ιταλίας και Κροατίας, Θέλω να πω ότι ενδιαφέρομαι πολύ να αξιολογήσω και να υποστηρίξω αυτή την Προεδρία, την Κροατική. Και να θέσω λοιπόν ίσως σήμερα την πιο επίκαιρη ερώτηση. Στα πλαίσια της ε, καθοδήγησής σας, πώς θα αξιολογούσατε τους κινδύνους στη Μεσόγειο από την πλευρά ασφαλείας, την κλιμάκωση ε, των εντάσεων που μπορούν να προκαλέσουν και άλλες μεταναστεύσεις και πολύ μεγάλη ανασφάλεια που θα είναι επιζήμια για την οικονομία μας όλα αυτά. Το Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα το θεωρείτε με αδιαφορία όπως η Φιλανδική Προεδρία ή θα δώσετε μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Κολακούσιτς έχει το λόγο. Πώς το ανήκει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε τη κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να θέσω κι εγώ με τη σειρά μου ένα ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε στην τρέχουσα κατάσταση που βλέπουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τους πιο σημαντικούς και μεγαλύτερους συνεισφορείς στον κοινοτικό προπολογισμό. Και ουσιαστικά καταβάλουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία λαμβάνουν ως δικαιούχοι. Η Κροατία από την άλλη είναι κυρίως χώρα δικαιούχος. Λαμβάνουμε περισσότερα κονδύλια από αυτά τα οποία συνεισφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ένας από τους πιο σημαντικούς συνεισφορείς προτίθεται να απαχωρήσει ενώ καταφθάνουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν ασταθείς οικονομίες και δεν πρόκειται με τη σειρά τους να συνεισφέρουν μεγάλα ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε επίσης και το λόγο ανάμεσα σε εργαζόμενο πληθυσμό και σταξιούχους. Στο παρελθόν, αυτό το οποίο είδαμε, ο λόγος αυτός ήταν τέσσερις εργαζόμενοι προς ένα σταξιούχο. Ενώ τώρα αν εξετάσουμε αυτή την αναλογία, στην Κροατία τουλάχιστον έχουμε 1,1 εργαζόμενο για ένα συνταξιούχο. Και βλέπω ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη. Δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή στην Κροατία και τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καταβάλουμε τις συντάξεις των μελλοντικών συνταξιούχων. Ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν εποφελούνται αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει καταβάλει πάνω από 150 δισεκατομμύρια, επιπλέον μάλλον, στον κοινοτικό προπολογισμό. Αλλά έχει, είχε ως απόδοση, ως κέρδος, 880 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, συνεισφέρουν σημαντικά, αλλά η απόδοσή τους είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να στηρίξουν χώρες με χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη σαν τη δική μας. Η στάση της κορατίας ποια θα είναι και ποιες είναι οι σχετικές δικές μας προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθότι θα είναι η τελευταία μου παρέμβαση, ελπίζω, στην ε, Επιτροπή αυτή, να σας δώσω κάποιες συμβουλές. Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit και τα σχετικά προβλήματα τα οποία τονίσαμε, τότε ε, ο πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε πει ότι η λύση ήταν περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Βέβαια, αυτό για μένα είναι πραγματικά κατανόητο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μέσω τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία έθιξε το Brexit. Στη δική μα Επιτροπή των Προπολογισμών, πολλοί ευρωβουλευτέ μα έχουν πει ότι καθότι τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν περισσότερα χρήματα από ό,τι είχαν πριν από μια δεκαετία, για παράδειγμα, θα πρέπει να συνεισφέρουν όλο και περισσότερο στο κοινωνικό προπολογισμό. Εγώ εκλέγομαι στην βορειοδυτική Αγγλία και υπάρχουν εκεί οικογένειε που έχουν βασικά προβλήματα βιοπορισμού. Το να ζητήσει κανεί από τι οικογένειε αυτέ ή από ανάλογε οικογένειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρουν περισσότερο στον κεντρικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώ ανεύθυνο. Ανταυτού, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξοικονομούμε στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού και να ταπανούμε περισσότερα κονδύλια. Όταν το 1972 προσχώρησε τότε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή, ε, στην ΕΟΚ μάλλον, τις χώρες ουσιαστικά σε μία αγορά. Αν ρωτούσαμε τους πολίτες στη Βόρεια Ευρώπη αν θέλουν πραγματικά μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή μία υπερευρώπη, θα σας λέγανε ότι προτιμούν το πρώτο. Ακριβώς αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιστρέψει στην κοινή ενιαία αγορά, να γίνει ουσιαστικά ένας χώρος ε, οικονομικών συναλλαγών, ελεύθερου εμπορίου και τίποτα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένω το Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει να προσχωρήσει εκ νέου στη νέα αυτή τότε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω άλλου ομιλητέ στον κατάλογο των αγορητών. Επομένω, να δώσω πολύ ευχαρίστω εκ νέου το λόγο στον Υπουργό, τον κύριο Μάριτς. Ακούσαμε, κύριε Υπουργέ, πολλές παρατηρήσεις, πολλές ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να σα ευχαριστήσω όλους που θέσατε ερωτήσεις, θίξατε διάφορα ζητήματα, κάνατε παρατηρήσεις, φωτίσατε διαφορετικές πτυχές του όλου ζητήματος. Εν τέλει πάντως, από προσωπικής τουλάχιστον πλευράς, πιστεύω ότι καταδείξατε το έντονο ενδιαφέρον αλλά και τις πολλές σχετικές ικανότητες και την περιογνωμοσύνη που έχετε για τα ζητήματα τα δημοσιονομικά. Όπως είπα στην αρχική μου παρέμβαση, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο στον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθότι όμως εφήγει όλος ιδιαίτερος το ζήτημα αυτό στις διάφορες ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας, θα προσπαθήσω να σας δώσω ακόμα περισσότερες πληροφορίες με τον κίνδυνο βέβαια να επαναλάβω κάποια στοιχεία τα οποία έθιξε ήδη στην αρχική μου παρέμβαση. Χαίρομαι πολύ που κι εσείς ε, αναγνωρίστε το ζήτημα αυτό ως πολύ σημαντικό και να σε ευχαριστήσω επίσης για την πολύ θερμή υποδοχή που επιφυλάξετε σε μένα και στην ομάδα μου. Ως κρατική Προεδρία θα θέλαμε προφανώς να έχουμε μια στενή και ισχυρή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο στον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις σχετικές διαπραγματεύσεις, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ενδιαφέρει την ε, δική σας την ε, Επιτροπή. Θεωρώ ότι η επικοδομητική αυτή σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως πολλά πράγματα στη ζωή και πολλά προβλήματα στη ζωή, έτσι και τα ζητήματα τα οποία θίξετε μπορούν να επιληθούν μέσω του διαλόγου. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε την ε, θετική αυτή πρακτική που ξεκίνησε στο παρελθόν κάθε φορά που θίγεται ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το πολιτέ στο πλαίσιο. Κάθε φορά που έχουμε νέε πληροφορίε, κάθε φορά που έχουμε νέε εξελίξει, θα είμαστε παρόντε για να συζητάμε και να ενημερώνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα πιο κρίσιμα στοιχεία του φακέλου αυτού, οι πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ που θα μα καθοδηγήσουν στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ένα από τα πολλά ζητήματα που εθίγησαν και το είπατε κι εσεί ήταν το είπε και ο αυτό, το ζήτημα των ιδίων πόρων και το ζήτημα της διοργανικής συμφωνίας. Όσον αφορά τους ε, ιδίους πόρους και όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, καθώς επίσης και κάποια άλλα ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης και αντικείμενο διαπραγματεύσεων στου τριμερούς διαλόγους. Αυτή τη στιγμή βέβαια εγκριθεί πρώτα η πολιτική καθοδήγηση. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους ίδιου πόρους, Ήδη είμαστε έτοιμοι γιατί η τεχνική εργασία στο Συμβούλιο έχει ήδη ολοκληρωθεί όσον αφορά το φάκελο αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν λάβουμε την πολιτική καθοδήγηση από το Συμβούλιο θα ξεκινήσουμε την ανάρθρο εξέταση των νομοθετικών προτάσεων που άπτονται του πακέτου των ιδίων πόρων. Θίξατε επίσης και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του μεγέθους του προπολογισμού. Αναφερθήκατε σε ποσοστά στην πρόταση την αρχική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην πρόταση που έκανε εν συνεχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα η τελευταία παρέμβαση που ακούσαμε ήταν λίγο διαφορετική. Μα είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερε εξοικονομήσει αντί να αυξάνουμε τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν εδώ πέρα ομοιότητες με την κατάρτιση του εθνικού προπολογισμού. Ανάλογες συζητήσει ή απόσταση απόψεων εκφράζεται και κατά τη διάρκεια του εθνικού προπολογισμού στο δικό μου το κοινοβούλιο, που άλλοι θέλουν αύξηση του προπολογισμού και άλλοι προτιμούν εξοικονόμηση. Προφανώ, στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού θα πρέπει να έχουμε έναν βιώσιμο προπολογισμό, ο οποίο να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και ρεαλιστικό και να συνάδει βέβαια με τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Οι δύο τελευταίε παρεμβάσει επικεντρώθηκαν περισσότερο στο Brexit. Προφανώ, η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική και δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Ο Ευρωβουλευτής κ. Κολάσιτς ε, έθεσε πολύ σωστά το ζήτημα τι θα γίνει με την απώλεια της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Brexit αποτελεί βέβαια γεγονός, επομένως θα πρέπει να το αποδεχθούμε και είμαι πεπισμένος ότι ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη αυτήν και θα δοθεί η απαραίτητη τελικά υποστήριξη προς τον κοινοτικό προπολογισμό κάτι το οποίο χρειαζόμαστε προκειμένου να καταφέρουμε να αποκριθούμε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πολύ σημαντικές προσδοκίες από εμάς και προφανώς εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Βέβαια, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών όχι μόνο μέσω του προπολογισμού αλλά και μέσω της νομοθεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επίσης όρει θα συζητήσουν ένα άλλο, με άλλη σημαντική νομοθετική πρόταση, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ξέρετε ότι κάναμε μια διεξοδική συζήτηση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και χθε το πρώτο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ κάναμε μια ανάλογη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συζήτηση ιδιαίτερα δυναμική και επικοδομητική, καθότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη συζήτησαν το ζήτημα αυτό και την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως Προεδρία, και αυτό ήταν και το μήνυμά μας προς το Συμβούλιο, και προς τα κράτη-μέλη, αλλά και προς εσάς, ότι ως Προεδρία θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, προκειμένου να διοργανώσουμε όλες τις απαραίτητες ε, συνεδριάσεις και τεχνικής φύσης στο επίπεδο του Συμβουλίου αλλά και αλλού, προκειμένου να προωθήσουμε τη συζήτηση και το διάλογο για την πολύ σημαντική νομοθετική αυτή πρόταση που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Νομίζω ότι ε, θα απαιτηθούν όχι μόνο μήνες, αλλά θα έλεγα ακόμα και χρόνια μέχρι να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το πλαίσιο διαπραγματεύσεων, το οποίο θίξατε ορισμένοι στις παρατηρήσεις σας, ο ρόλος εδώ του Ευρωπαϊκού Συνοβουλίου συνάδει με το ρόλο που προβλέπετε γι' αυτό από τις συνθήκες. Θα πρέπει να δώσουμε εμεί την απαραίτητη όθηση και να καταφέρουμε να δώσουμε την απαραίτητη πολιτική καθοδήγηση και τι απαραίτητε πολιτικέ προτεραιότητε. Η πολιτική λοιπόν αυτή καθοδήγηση που θα δοθεί από το ανώτατο επίπεδο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την στασιμότητα, την τελμάτωση αυτή στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πάντως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητε προϋποθέσεις προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος και σε αυτό θα συμβάλλει βέβαια και η πολιτική καθοδήγηση που περιμένουμε από το Συμβούλιο. Και βέβαια, όπως ε, σας είπα και πριν από λίγο, εμείς θα είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε την όλη συζήτηση. Ορισμένοι θίξατε το ζήτημα των αιτήσεων προπολογισμών και συγκεκριμένα του προπολογισμού για το 2021. Και ως προς αυτό το Συμβούλιο προετοιμάζει αυτή τη στιγμή την πολιτική του καθοδήγηση για τον αιτήσιο αυτό προπολογισμό. Η πολιτική αυτή καθοδήγηση θα παρουσιαστούν στους αρμοδίους εκπροσώπους των κρατών μελών την Άνοιξη και αυτή τη στιγμή υποβάλλει το προσχέδιο προπολογισμού Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, θα είναι η επερχόμενη Γερμανική Προεδρία που θα ηγηθεί τη όλη διαδικασία. Ορισμένοι θίξατε το ζήτημα του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε την δυναμικότητα ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και των μεμονωμένων κρατών μελών. Και θα αναφερθώ και στα όσα θίξατε όσον αφορά τις δημογραφικές στάσεις και τη μετανάστευση. Πάντως, ένα από τα μέσα, ένα από τα εργαλεία που έχουμε προκειμένου να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ελκυστική είναι το μέσο αυτό της ε, στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Το ίδιο ισχύει και για του ιδίου σπόρου. Πάλι και εδώ περιμένουμε μια πολιτική καθοδήγηση και αυτή τη στιγμή θα την έχουμε θα καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερου διαπραγματεύσει. Πάντω, όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξη των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συμφωνήσουμε όπω είπατε και επί τη μεθοδολογία και τη ορολογία που ακολουθεί το Συμβούλιο. Ω προ αυτό θα έχουμε μια μερική γενική προσέγγιση στο πρώτο τρίμηνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έχουμε την πολιτική καθοδήγηση όπως σας είπα. Θα αρχίσουμε να συζητάμε το πρόγραμμα αυτό στηρίξη των μεταρρυθμίσεων. Αναφέρατε και ένα ακόμα ζήτημα βέβαια. Το ζήτημα της μετανάστευσης. Προφανώς αναφέρομαι στην ε, Κροατία και πλέον μιλάω ως υπουργό Οικονομικών της Κορατίας και ως εκπρόσωπος της κορατικής κυβέρνησης και όχι ως εκπρόσωπος της κορατικής προεδρίας. Εξ αρχής, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή η προσφυγική μεταναστευτική κρίση, η στάση της Κορατίας ήταν σαφής και ξεκάθαρη και ιδιαίτερα διαφανής. Είχαμε εξ αρχής πει ότι θα αναλάβουμε δυναμικά δράση για τη διαχείριση των συνόρων μας, Μολονότι βέβαια η Κροατία δεν είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, 56.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχει έκταση. Ακριβώς όμως επειδή έχει την ιδιαίτερη αυτή ε, μορφολογία και σχήμα, έχει πολύ σημαντικά εκτεταμένα εξωτερικά σύνορα με όλες τις γειτονικές χώρες και ιδίως με την Βοσνία Ερζεγοβίνη σύνορα στα οποία τώρα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Εγώ νομίζω ότι ε, τα πάμε καλά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξει τελικά σε μια θετική αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ε, τα θεσμικά μας όργανα χειρίζονται τα εξωτερικά μας σύνορα. Ακολουθούμε συγκεκριμένα πρότυπα, μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και νομίζω ότι η θετική αυτή αξιολόγηση που θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελέσει την καλύτερη δυνατή απόδειξη ότι τα πράγματα κινούνται θετικά και όπως ξέρετε θέλουμε σύντομα να ενταχθούμε και στο χώρο Σέγγεν. Εξ αρχής πάντως από τότε που ξέσπασε η μεταναστευτική κρίση είχαμε πει ότι θα αναλαμβάναμε μια αποτελεσματική δυναμική δράση και ότι θα παρήχαμε σε όλους τους πρόσφυγες την απαραίτητη στέγαση αλλά και τις απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες. Σίγουρα όμως αντιμετωπίζουμε δύσκολες προκλήσεις και όπως θα έχετε δει ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και η Ιταλία αλλά και άλλες μεσογειακές χώρες. Ανάλογα προβλήματα και προκλήσεις λοιπόν αντιμετωπίζουμε και εμείς και βέβαια χρειαζόμαστε μια συλλογική προσέγγιση καθώς επίσης και την κατανόηση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι η Κροατία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται δυναμικά και ενεργά την όλη αυτή κατάσταση και ένα πολύ μεγάλο μέρος των πόρων μας κατευθύνεται ήδη προς την διαχείριση αυτή των εξωτερικών μας συνόρων. Να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και αυτό με τη μετανάστευση και θα αναφερθώ στις δημογραφικές τάσεις. Ως Κροατική Προεδρία Ήδη έχουμε θέσει το ζήτημα αυτό στις προτεραιότητές μας και σε διάφορα φόρα επίσης θα το θέσουμε εκ νέου και στο Συμβούλιο Κοφίν, για παράδειγμα, στην άτυπη συνεδρίαση που θα γίνει στο Ζάγκρεπ στις 24 και 25 Απριλίου θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της δημογραφίας, των δημογραφικών τάσεων και βέβαια εδώ δεν θα συζητήσουμε μόνο τις μεταναστευτικές προκλήσεις και την εσωτερική μετανάστευση, αλλά και τις γενικότερες δημογραφικές τάσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας περιέγραψα λίγο την κατάσταση της Κροατίας. Ακούσατε από έναν ε, Ευρωβουλευτή ποια είναι η αναλογία μεταξύ ενεργού πληθυσμού και συνταξιούχων. Αναφερόμαστε βέβαια εδώ πέρα σε διάφορα συστήματα τα οποία επηρεάζονται, το εξαιρετικό σύστημα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το σύστημα δημόσιας υγείας. Κάθε χώρα πάντως, κάθε εθνικό σύστημα, κάθε κοινωνία επηρεάζεται διαφορετικά από τα ζητήματα αυτά, αλλά και πάλι το θέμα θεωρώ ότι είναι σφαιρικό και συλλογικό. Δεν νομίζω ότι ε, Υπάρχουν συνάδελφοι υπουργοί που να μην γνωρίζουν τελικά ότι οι προκλήσεις αυτές μας αφορούν όλους και ότι είναι ιδιαίτερα αναδυόμενο στο τελευταίο διάστημα και θα πρέπει να βρούμε κάποιε συλλογικέ λύσει. Οτιδήποτε κάνουμε λοιπόν σε σχέση με τι προτεραιότητε των μεταρρυθμίσεων, είτε πρόκειται για το σύστημα δημόσια υγεία ή το σύστημα κοινωνική ασφάλιση ή το ζήτημα το σταξιδοτικό, δεν υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει μία ενιαία μαγική λύση. Αυτό το οποίο αποτείται λοιπόν είναι να έχουμε μία υγιή, ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη που θα δημιουργήσει απασχόληση, θέσεις εργασίας. Και σε σχέση με την ερώτηση που έθεσε ο Ευρωβουλευτή για την αναλογία μεταξύ εργαζόμενου πληθυσμού και συνταξιούχων, μία θα μπορούσε να βρεθεί από αυτό. Νομίζω ότι είναι απλά μαθηματικά, έτσι δεν είναι. Αριθμητής και παρονομαστής. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο θίξατε. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Ελπίζω ότι και εσείς αποτιμάτε ως ιδιαίτερα θετική τη σημερινή μας συζήτηση. Έχω καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις σας, όλα τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Πραγματικά εμπλουτίσατε τη συζήτηση με πολλέ νέε ιδέε, φωτίσετε πολλέ διαφορετικέ πτυχέ όλων αυτών των ζητημάτων και σα διαβεβαιώ ότι η Κροατική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες της στο επίπεδο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα προωθήσουμε βέβαια και τον διάλογο και τον συντονισμό και με εσά για αυτό το ζήτημα και για πολλά άλλα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμεί σα ευχαριστούμε κυρία Μάριτ για την διεξοδικότατη απάντηση στα σχόλιά σα ε, για τι διάφορε παρατηρήσει των συναδέλφων μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για το ότι ήσασταν εδώ πρώτα απ' όλα και ελπίζω να ξαναέλθετε στο μέλλον. Είστε καλοδεχούμενος. Σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν και πάρα πολύ ειλικρινείς και ανοιχτός απαντής σας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ομάδα μας. Και μια και σας έχουμε εδώ, δεν θα σας αφήσουμε γιατί ξέρετε ότι θα είμαστε τη Δευτέρα στο Ζάγκρεπ με τη θερματιστική ομάδα για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Οπότε θα σας ξαναδούμε εκεί με μεγάλη χαρά. Θα ε, ξανασυνεδριάσουμε στις 3 το μεσημέρι.